Uh, Αγαπητοί μου φίλοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη εισαγωγή. Uh, δεν ήταν δική μου ιδέα να, ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε τη συνεδρία στις 2.30. Προτιμώ η μεσημεριανή διακοπή, η σχέστα μας να είναι πιο παρατεταμένη. Παρόλο που δεν είμαι ούτε από την Ιταλία ούτε την Ισπανία, μου αρέσει η τα. Πάντως χαίρομαι που μερικοί από εσά ε, δώσατε το παρόν και τόσο νωρί. Γιατί πρώτο σημείο της απογευματινή ημερήσιας διαταξη είναι η δεύτερη μα συνάντηση, γιατί η πρώτη συνάντηση με την Επίτροπο ήταν η ακρόασή τη. Έχουμε τώρα τη δεύτερη συνάντηση, πολύ σημαντική, γιατί στην Επιτροπή μας ε, νιώθουμε υπεύθυνοι για την ψηφιακή ένωση. Όχι τόσο για την ενία ψηφιακή αγορά, για πραγματική ψηφιακή ένωση. Οπότε, όταν βλέπετε ανταλλαγή απόψε με την Επίτροπο για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, για θέματα του πακέτου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και την ελεύθερη κυκλοφορία των μη προσωπικών δεδομένων ως τμήμα του διαρθρωμένου μας διαλόγου, καταλαβαίνετε ότι η συζήτηση θα είναι πολύ σημαντική. Και επίσης ε, έχουμε το κοινό μας πρόγραμμα το 2018 που περιλαμβάνει ε, την πρόταση για τον Μπερεκ, ε, τον Οργανισμό Συντονισμού Ελεκτρονικών Επικοινωνιών. Οπότε βρισκόμαστε στα μέσα της διαδικασίας και για το θέμα του ΜΠΕΡΕΚ και να επισημάνω ότι εγκρίναμε και την έκθεσή μας για την Ομάδα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Τηλεπικοινωνίες, τον ΜΠΕΡΕΚ, μόλις την περασμένη εβδομάδα και οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο αναμένεται να ξεκινήσουν ως ονούπο. Οπότε είμαστε έτοιμοι για τον τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο για, το, για τον κώδικα ηλεκτρονικών ε, επικοινωνιών και την πρόταση για το Φορέ Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τον ΠΕΡΕΚ δηλαδή. Και τώρα θα εξετάσουμε ε, το πακέτο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την ελεύθερη ροή μη προσωπικών δεδομένων. Γιατί είναι θέματα δικής μας αρμοδιότητα, συναρμοδιότητα μάλλον, με την Επιτροπή ε, Εσωτερικής Αγοράς και προστασία των Καταναλωτών, γιατί είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους καταναλωτές μας. Παρακαλώ κυρία Επίτροπε, έρχεται το λόγο για την ε, εισαγωγική σα ομιλία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπούζεκ. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, καταρχήν σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να καταστήσουμε πραγματικότητα την ενιαία ψηφιακή αγορά που επηρεάζει την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι πολύ σημαντικό θέμα και ψυχοτικό, βλέποντας με τι γοργό ρυθμό προχωρεί η Επιτροπή σας στα θέματα της ψηφιοποίησης. Γιατί γνωρίζετε όπως και εγώ ότι αυτή η ενιαία ψηφιακή αγορά ξεκίνησε σε ένα πλαίσιο. Είναι μία από τις δέκα προτεραιότητες της παρούσας επιτροπής ε, με τον πρόεδρο τον Ζαν ε, Γιουνκέρ. Έχουμε 24 προτάσεις επιτάπητος, 6 έχουν ολοκληρωθεί. 18 προτάσεις απομένουν και για αυτές θα πρέπει να συνεργαστούμε για να τις διεκπαιρεώσουμε αισίως μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους και μακάρι και λίγο νωρίτερα. Όλες αυτές οι προτεραιότητες άλλωστε καθορίστηκαν και χαρακτηρίστηκαν ως προτεραιότητες και από τους τρεις Προέδρους. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό επιτρέψτε μου να επιστήσω την προσοχή σας σε τρία περιστατικά. Είχαμε αφενός ε, την ε, διάσκεψη κορυφής ε, των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στο Τάλιν πριν από δέκα μέρες. Ήταν καθοριστική αυτή η διάσκεψη κορυφής γιατί ε, έδωσε ένα ακλόνητο και σαφές μήνυμα ότι η οικονομία μας, η απασχόλησή μας, οι πολίτες μας ζητούν διακαώς μια ενιαία ψηφιακή αγορά και μάλιστα πάρα αυτά. Αυτό το μήνυμα λοιπόν ε, θα ε, επαναληφθεί και επίσημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας και από την επόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί στο έκτακτο Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών της 24ης Οκτωβρίου. Χαίρομαι λοιπόν γιατί ε, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και από τους πολιτικούς μας ηθήνοντες ε, ε, διαπιστώθηκε επίγνωση αυτής της σημασίας ε, που έχει ψηφιακή αγορά. Θα ήθελα λοιπόν να επικεντρωθώ σε μερικές από αυτές τις προτάσεις. Καταρχήν, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Κυβερνοασφάλεια είναι η πιο πρόσφατη μας πρόταση από το 2013 όμως γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δική της στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Βέβαια, ο ρυθμός, η περιπλοκότητα και το εύρος των κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και οι συνέπειές τους στην κοινωνία και την οικονομία, αναπτύσσονται και μάλιστα με ανησυχητικούς ρυθμούς. Στόχος των μέτρων που προτείναμε είναι να συμβάλλει στην προστασία των πολιτών μας, των επιχειρήσεών μας και των δημοσίων φορέων και να τους θωρακίσει απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις και τις υβριδικές απειλές. Η πρότασή μας απορτίζεται από πολλά κέρια σημεία. Καταρχήν, από ένα κανονισμό που ανανεώνει την εντολή του Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. Ε, στόχος μας είναι να εφοδιάσουμε τον οργανισμό αυτό την ενίσα με μια πραγματική ικανότητα να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος ο οργανισμός αυτός ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών πρέπει να ε, ισχυροποιηθεί και να γίνει πιο αποτελεσματικός ώστε να μπορέσει να εφαρμόσει την ε, οδηγία νης από το 2016. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η δημιουργία ενός πλαισίου για την πιστοποίηση σε θέματα ασφάλειας των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Στόχος μας είναι να φροντίσουμε να μεριμνήσουμε ώστε τα προϊόντα και οι υπηρεσίες στην Ευρώπη και κυρίως ε, η εξάπλωση του διαδικτύου του διαδικτύου των πραγμάτων να ανταποκρίνεται στους κανόνες και τις προδιαγραφές μας για την κυβερνοασφάλεια. Επίσης, συντονισμός ώστε σε περίπτωση μιζώνων ε, περιστατικών επιθέσεων, ε, κυβερνοεπιθέσεων που επηρεάζουν πολλά μέτρα να έχουμε άμεση δράση. Γι' αυτό έχουμε και σχετική σύσταση και το πακέτο μας προ... περιλαμβάνει και σύσταση προς τα κράτη-μέλη να θέσουν σε εφαρμογή με αποτελεσματικό τρόπο την οδηγία νης. Ένα άλλο σημείο που μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές είναι η πρόταση για την ε, σύσταση ενός δικτύου ε, δεξιοτήτων και έρευνα σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις τεχνολογικές ικανότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Οπότε αυτά τα μέτρα θέλουν να εμπλέξουν όλους τους ενδιαφερομένους στον αγώνα αυτό και να το συντονίσουν και θέλω να υπολογίζω στη δική σας υποστήριξη ώστε να δώσουμε σάρκα και οστά σε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία. Ε, δεύτερο σημείο, ε, η ελεύθερη διακίνηση των δεδομένων, ελεύθερη ροή των δεδομένων. Ε, λαμβάνω ιδιαίτερα στα σοβαρά την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μεριμνήσει για την ελευθερία κυκλοφορίας προς των τεσσάρων ελευθεριών. Δεν μπορούμε λοιπόν να αναγκάζουμε τις επιχειρήσεις και τους ε, πολίτες ε, να κρατούν και να επεξεργάζονται τα δικαιώματα μόνο στην επικράτειά τους, εκτός ε, αν υπάρχουν πραγματικοί λόγοι δημόσιας ασφάλειας. Η... Τα εμπόδια στην ροή των δεδομένων δημιουργεί προσκόμματα και επιβαρύνει οικονομικά τις τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να αποφεύγουμε και επικαλύψεις σε θέματα πόρων πληροφορικής. Επίσης, μαζί με τους αυστηρούς κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων, ε, θα εφαρμόσουμε αυτή την πρόταση. Άλλωστε, ο κανονισμός GDPR προβλέπει ήδη την ελεύθερη ροή δεδομένων, προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα πρόταση εξασφαλίζει την ίδια κινητικότητα των δεδομένων για τα δεδομένα που δεν έχουν προσωπικό χαρακτήρα. Και η πρόταση είναι απλούστατη. Θεσπίζουμε κάποιε αρχέ για την ελεύθερη κυκλοφορία των μη προσωπικών δεδομένων και την διαθεσιμότητα των δεδομένων αυτών για τους δημόσιους φορείς, τι δημόσιε αρχέ. Εναπόκειται μετά στι δημόσιε διοικήσεις των κρατών μελών να εφαρμόσω την πρόταση. Βέβαια, οι στόχοι τη πρότασή μα ε, θα εφαρμοστούν και θα υλοποιηθούν πλήρω μόνο με συνεργασία με τα κράτη-μέλη και γι' αυτό προτείνουμε την ε, δημιουργία ενιαίων σημείων επαφής σε όλα τα κράτη-μέλη για να εξασφαλίσουμε ε, την άρση της υποχρέωσης ε, της αδικαιολόγητης τοποθέτησης, καθώς και την εφαρμογή, την έμπρακτη εφαρμογή του κανονισμού. Θα πρέπει να στηρίξουμε την ελεύθερη κίνηση των δεδομένων με συστήματα πληροφορικής, όταν οι επιχειρήσεις θέλουν να αλλάξουν παρόχους υπηρεσιών, για παράδειγμα. Ε, με την πρότασή μας θα φροντίσουμε ώστε αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών να αναπτύσσουν κώδικες αυτορύθμισης για να διευκολύνουν τις αλλαγές. Τρίτο θέμα αφορά μετά το B2B και το B2C έχουμε το P2B, δηλαδή στις σχέσεις ιδιωτών επιχειρήσεων. Το ψηφιακό μας έργο και τα ψηφιακά μας καθήκοντα δεν σταματούν εδώ. Θα έχετε εντός ολίγου κάποια μέτρα που στόχο έχουν την ε, καταπολέμηση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών που έχουν εντοπιστεί μεταξύ των επιχειρήσεων που διαδικτυακά διαθέτουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους και των παρόχων αυτών των, των πλατφορμών. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ισότιμους ε, όρους ανταγωνισμού και θεμητού ανταγωνισμού, ώστε να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να έχουμε έναν υγιή τομέα ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη. Τέταρτο θέμα, κώδικας ε, ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το θέμα δηλαδή για το οποίο ε, η Επιτροπή σας, η Ήτρε, έπαιξε και θα συνεχίσει να παίζει σημαντικό ρόλο. Καταρχήν να συγχαρώ την κυρία Πιλάρ Καστίγιο, την εισηγήτριά σας, για την έγκριση του σχεδίου έκθεσή της και συγχαρητήρια για την την χαρμόσυνη είδηση στην προσωπική της ζωή. Επίσης, ε, κάτι τέτοιο θα γίνει μόνο αν έχουμε ένα προβλέψιμο πλαίσιο που θα δίνει κίνητρα στους ε, τελεστές για επενδύσεις. Χαίρομαι που εγκρίνατε τα, τις περισσότερες προτάσεις μας για το φάσμα και κυρίως την ανάγκη ενός συντονισμένου χρονοδιαγράμματος ε, των κατανομών και την, τα 25 χρόνια για τη διάρκεια των αδειών εκμετάλλευσης του φάσματος. Κάτι τέτοιο είναι σημαντικό για την κινητή διασυνδεσιμότητα. Και φυσικά λαμβάνω υπόψη την ρήτρα ενδιάμεση αξιολόγηση που συμπεριλάβατε και στις μελλοντικέ διαπραγματεύσεις ε, ε, θα προσέξω ιδιαίτερα αυτό το θέμα της διάρκειας γιατί είναι πολύ σημαντική για την προβλεψιμότητα των επενδύσεων. Επίσης, ε, για τις επενδύσεις είναι σκόπιμο για τους επενδυτές να μπορούν να προβλέπουν αν θα υπάρχει ρύθμιση για ένα δίκτυο ή όχι. Και χαίρομαι που αντισταθήκατε στο αίτημα να ε, επεκτείνουμε σε όλους τους παρόχους την υποχρέωση πρόσβασης σε δίκτυα μεγάλης ικανότητας, άσχετα με την ισχύ τους στην αγορά ε, δηλαδή την επιβολή ε, συμμετρικών υποχρεώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρόταση λιγότερο άκαπτης νομοθεσίας καινοτόμησε και έτσι διευκολύνει την ανάπτυξη δικτύων ε, μεγάλης ε, ταχύτητας, μεγάλης ικανότητας. Οπότε, αν οι ε, συμμετέχουν σε αυτό το κόστος ανάπτυξης, θα βοηθήσουν στην κάλυψη μεγαλύτερων γεωγραφικών ζωνών που θα έμεναν εγκαταλελειμμένες οι δεμοί. Βέβαια, έχω υπόψη την ανάγκη να μην γίνουν όλα αυτά εις βάρος του, του ανταγωνισμού. Θα πρέπει να θεσπιστούν οι απαραίτητε ασφαλιστικές δικλείδες. Πάντως, τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τα κανονιστικά μέτρα να είναι σαφή από την αρχή. Διαπιστώνω ότι η Επιτροπή σας δεν συμφωνεί με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεωρεί ότι μια ρύθμιση θα πρέπει να περιορίζεται στο να επιλύει τα προβλήματα σε επίπεδο τελικού καταναλωτή ή λιανικού εμπορίου, λιανικής αγοράς. Ελπίζω όμως ότι θα συμφωνήσουμε τελικά ως προς την αρχή ότι η ρύθμιση θα πρέπει να λύνει τα προβλήματα της πραγματικότητας και θα πρέπει από τον ανταγωνισμό να επωφελούνται όλοι αλλά να μπορούν και να αναπτύσσονται σε περίπτωση που οι συνθήκη τη αγορά είναι ανεπαρκεί. Θα πρέπει να καθησυχάσουμε του επενδυτέ ότι δαπανηρέ επενδύσεις δεν θα υποβάλλονται σε περιττή ε, νομοθετική ρύθμιση. Σε ό,τι αφορά τον Μπερέκ, ε, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Τοσενόφσκι, τον εισηγητή σας, για το έργο που επιτέλεσε ως προς ε, τον την έκθεση για το Φορέα Ευρωπαϊκών Ερυθμιστικών Αρχών. Αν θέλουμε μία πρόταση που θα δράσει σε αρχές, θέλουμε έναν ε, μηχανισμό αποτελεσματικής, αποτελεσματικού συντονισμού και μία αποτελεσματική διακυβέρνηση. Ε, συμφωνώ λοιπόν με την πρότασή σας και λυπάμαι μάλλον που εσείς δεν συμφωνείτε με, τη, το σχηματισμό του ΜΠΕΡΕΚ σε ένα ε, πλήρη φορέα και ευρωπαϊκό οργανισμό με, δημοκρα... με διοικητικό συμβούλιο. Αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να καταστήσουμε τον ΜΠΕΡΕΚ πιο υπεύθυνο και αποτελεσματικό και να το εφοδιάσουμε με μια ε, νομική ε, προσωπικότητα. Η ευθύνη και η διαφάνεια είναι απαραίτητες για να ενισχυθεί ο ρόλος του φορέα ΜΠΕΡΕΚ σε θέματα ρύθμισης. Λαμβάνω υπόψη τις ανησυχίες σας για την ανεξαρτησία του Μπερέκ που ενδεχομένως διακυβευτεί από τη συμμετοχή στην ψηφοφορία της Επιτροπής στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο και την επιλογή του εκτελεστικού διευθυντή. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να υπονομεύσουμε, να υποσκάψουμε την ανεξαρτησία του Μπερέκ. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σα για να διασκεδάσουμε τι ανησυχίε σα. Και για έναν ισχυρό φορέα Μπερέκ, η επιλογή του συνόλου των αριθμιστών, μεγάλων και μικρών, θα πρέπει ε, όλε οι φωνέ να έχουν την ίδια αξία και βαρύτητα. Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό αν το τεχνικό έργο. Ε, δεν ρυθμίζεται παρά μόνο από τους μεγάλους που είναι οι καλύτερα εξοπλισμένοι ρυθμιστές. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας και κυρίως τον εισηγητή τον κύριο Σοχίνιο για μια πρωτοβουλία που μου είναι ιδιαίτερη, ιδιαίτερα προσφυλής, το Wi-Fi for EU. Και χαιρετίζω το έργο σας ως προς τον γεωγραφικό αποκλεισμό Μπράβο στην κυρία Κάλλη, Καηλή, στην οδηγία κύριε Κρασοντεύσκη χαρητήρια και στον κανονισμό κυρία Μλινάρ ε, και για τα πνευματικά δικαιώματα και τον κανονισμό για την ηλεκτρονική ιδιωτική σφαίρα, το e-privacy της κυρίας Κάλλα. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Αυτά εισαγωγικά και περιμένω τη συζήτηση και τις ερωτήσεις σας, ε, στις οποίες ελπίζω ότι θα απαντήσω με ικανοποιητικό τρόπο. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την εισαγωγική σας αυτή παρέμβαση στην αρχή της ε, συζήτησης. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους που είναι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων να πάρουν τώρα το λόγο. Πρώτος ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την ξεκάθαρη αυτή παρουσίαση. Θέσατε συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους πρέπει να πετύχουμε. Είναι οι στόχοι που έχουμε θέσει τώρα το φθινόπωρο του 2017 και θεωρώ ότι μέχρι του χρόνου το φθινόπωρο θα πρέπει να εργαστούμε πάρα πολύ σκληρά προκειμένου να επιτύχουμε όλους αυτούς τους στόχους που έχουν να κάνουν με την ψηφιακή ενιαία αγορά. Θα ήθελα να σας θέσω ερωτήματα σχετικά με κάποια ζητήματα. Πρώτον, Πώς αξιολογείτε εσείς την κατάσταση όσον αφορά την εργασία που γίνεται για τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ελεκτρονικών Επικοινωνίων. Πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε πάρα πολύ στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου. Πρέπει να καταλήξουμε γρήγορα σε ένα συμπέρασμα, σε μια απόφαση. Και έπειτα όσον αφορά τη διαχείριση και την κατανομή του φάσματος και προς αυτό τι έχει να μας πείτε. Έπειτα τα ζητήματα που άπτονται της κυβερνοασφάλειας. Ποια είναι η δική σας άποψη κύριε Επίτροπε. Πιστεύετε ότι χρειάζεται μια πιο ισχυρή συνεργασία και ένας πιο έντονος συντονισμός και μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με τα ζητήματα κυβερνοασφάλειας και είναι δυνατό κάτι τέτοιο ή θα καταλήξουμε στην ίδια κατάσταση με αυτή που αντιμετωπίζαμε και αντιμετωπίζουμε ακόμα κάθε φορά που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε την οδηγία όσον αφορά την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών όπου βλέπουμε ότι προκύπτουν πολλές καθυστερήσεις και πολλά προβλήματα σε πολλές χώρες και όσον αφορά πάλι τα ζητήματα κυβερνοασφάλειας Ποια είναι η άποψή σα όσον αφορά τα συστήματα πιστοποίηση. Ξέρετε ότι ε, όταν ασχολούμεθα με το διαδίκτυο των πραγμάτων, το σύστημα αυτό πιστοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη όμω πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε μία ενιαία μόνο λύση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να καλύπτει όλε τι περιπτώσει. Πρέπει να δούμε πώ μπορεί το σύστημα αυτό πιστοποίηση να καλύψει όλου του οικονομικού τομεί και πώ μπορούμε να εμπλέξουμε όλου του οικονομικού και βιομηχανικού τομεί. Και μια τελευταία ερώτηση με την αδειά σας κύριε Επίτροπε όσον αφορά την έντολή της ΕΝΗΣΑ. Αναφερθήκαμε στι νέε αρμοδιότητε που θα έχει ο Οργανισμό Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών σε σχέση με την κυβερνοασφάλεια για την προστασία των ίδιων των πολιτών. Από την άλλη όμως θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων των πολιτών και θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και διεθνών οργανισμών όπως το ΝΑΤΟ. Θα αξιολογήσετε λοιπόν και τη δυνατότητα αυτή προκειμένου να υπάρχουν κάποια κοινά προγράμματα, προγράμματα κατάρτισης, γιατί νομίζω θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ιδίως για ζητήματα κυβερνοασφάλειας. σε ευχαριστούμε πολύ. Εξ ονόματος τώρα του ECR, ο κύριος Τοσενόφσκι έχει το λόγο κύριος Νίλκαν, συγγνώμη, ο κύριος Τσοτινόφσκι μόλις έφτασε και γι' αυτό αναφέρθηκα σε αυτόν. Ο κύριος Νίκα, εξ ονόματος των σοσιαλιστών. Σας το συγγνώμη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Συνειδητοποιώ ότι πήρατε το λόγο για ζητήματα τα οποία είναι αρκετά πολύπλοκα και χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε πάλι σύντομα να μας δείτε. Ο Επίτροπος Έτιγκερ έκανε πρόσφατα μία αναφορά στο ζήτημα της κοινή λογικής που θα πρέπει να πριτανεύσει όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο τόσο για τους καταναλωτέ του πολίτε ω και τι επιχειρήσει, Ασφάλεια όσον αφορά τα συστήματα πληροφορική. Νομίζω ότι εδώ πέρα θα μπορούσαμε να είχαμε ένα είδο βαθμολόγηση τη ποιότητα, όπω γίνεται για παράδειγμα στον τουριστικό τομέα για τα ξενοδοχεία. Ο κύριο Σέτιγκερ πρότεινε να υπάρχει ένα αντίστοιχο σύστημα και μια αντίστοιχη βαθμολόγηση όσον αφορά την ασφάλεια στο διαδίκτυο και ουσιαστικά να επιβραβεύουμε αυτού οι οποίοι επενδύουν σε συστήματα τα οποία είναι ασφαλή και κατά αυτόν τον τρόπο θα στείλουμε και ένα ηχηρό μήνυμα και προς τους καταναλωτές και γενικότερα προς τους πολίτες για τις συσκευές εκείνες ή τα προγράμματα εκείνα τα οποία δεν αναγνωρίζονται και δεν πιστοποιούνται ως ποιοτικά ή ασφαλή στον κυβερνοχώρο. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή διστάζουν ορισμένοι να κάνουν τι απαιτούμενε επενδύσει στο ζήτημα τη ασφάλεια του κυβερνοχώρου και δυστυχώ ε, αυτό δεν βοηθά ιδιαίτερα τους καταναλωτές, οι οποίοι καλούνται αυτή τη στιγμή να επιλέξουν ανάμεσα σε σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες και δεν ξέρουμε τελικά αν ε, θα επιλεγούν περισσότερο προϊόντα υπηρεσίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τις ΗΠΑ και πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα δεν έχουν κινηθεί καθόλου όσον αφορά την ε, εξέλιξη των ασφαλών υπηρεσιών στα πλαίσια του κυβερνοχώρου, αλλά ακόμα και στα πλαίσια της διοίκησης του ναυτή χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες οι οποίοι στην καθημερινότητά τους φοβούνται, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουν διαδικτυακά τραπεζικά συστήματα, φοβούνται ότι μπορούν να χάσουν κατά αυτόν τον τρόπο τα χρήματά τους. Νομίζω ότι ο κύριος Έτιγκερ σε όλα αυτά τα ζητήματα αναφερόταν όταν έκανε λόγο για βαθμολόγηση και επιστοποίηση προγραμμάτων. Ξέρετε ότι υπάρχουν διάφορα προγράμματα τα οποία οι εφαρμογέ που μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τηλεφωνικά μα δεδομένα ή σε φωτογραφίε μα ακόμα και προσωπικέ ή σε πολλά άλλα προσωπικά ή οικονομικά δεδομένα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θέτει ένα τεράστιο πρόβλημα ασφάλεια. Με... Ξέρω ότι μπορεί να λάβει κανεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ουσιαστικά να απαιτεί από τον παραλήπτη να του δώσει πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά του δεδομένα. Τίθεται έπειτα και το ζήτημα της ε, ενίσα, της πιστοποίησης, των διασφαλίσεων. Νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία είπατε θα αποτελέσουν σίγουρα μια πολύ θετική εξέλιξη για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Όσοι επενδύσουν ουσιαστικά στον τομέα αυτό θα διαφοροποιηθούν ποιοτικά από τους υπόλοιπους. Ιδίως όσον αφορά το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας και νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς οι προτάσεις αυτές μπορούν να λειτουργήσουν στην πράξη και θα πρέπει να έχουμε και ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίηση σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων. Κυβερνοεπιθέσεις, οποίες βλέπουμε να πολλαπλασιάζονται όλο και περισσότερο. Ξέρετε ότι οι κυβερνοεπιθέσεις αυτές δεν απασχολούν ποτέ μόνο ένα κράτος μέλος ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης θα μπορούσε να προστατεύσει και πολλά άλλα κράτη-μέλη σε περίπτωση που έχουμε μια πρώτη επίθεση σε ένα κράτος. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται ένα, ένα τέτοιο σύστημα. Επίτα όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Θα πρέπει να δούμε πάλι εδώ πέρα ποιες θετικές εξελίξεις έχουμε, ποια είναι τα θετικά παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποια συστήματα τα οποία στρέφονται κατά των κακόβουλων ιών και ουσιαστικά μας προστατεύουν επίσης και από την κατάχρηση που μπορεί να γίνει ορισμένων συστημάτων στο διαδίκτυο. πιστεύω ότι θα μπορούσαν τέτοια μέτρα να χρησιμοποιηθούν και στα πλαίσια τη ε, ευρωπαϊκή αγορά προκειμένου να αυξηθεί η κυβερνοασφάλεια. Αναμένουμε περισσότερα ω προ αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλή επιτυχία σα εύχομαι πάντω. Uh, σα ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σα. Να ακούσουμε τον κύριο Τσοβανόφσκι από το ECR τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καταρχάς θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί καθυστέρησα. Ήταν δύσκολη η συνεδρίαση και ήταν και δύσκολες οι διαπραγματεύσεις με τους κοιότητες συζητητές για θέματα της ενέργειας. Και όλοι θα ξέρετε ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές ποτέ δεν είναι απλές, αλλά εν πάση περιπτώσει με ενημέρωσαν για την εισαγωγική σας ομιλία. Θα ήθελα λοιπόν να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την ε, προσέγγιση που ακολουθείτε στο θέμα αυτό σε ό,τι αφορά την όλη ψηφιακή τεχνολογία. Και έχω μία ερώτηση. Προετοιμάζοντας τις νομοθετικές προτάσεις για την ΠΕΡΕΚ και για τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ελεκτρονικών Επικοινωνιών με την συνάδελφο κυρία Δικαστήγιο, Ακούσαμε σε πολλές περιπτώσεις ερωτήσεις σε ό,τι αφορά την πτυχή της ασφάλειας και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Υπάρχει φυσικά ο οργανισμός και το ΜΠΕΡΕΚ. Θα ήθελα να αναφέρω όμως και το GSA. Μια υπηρεσία που βρίσκεται σε κίνδυνο το GSA λοιπόν πιστεύω ότι έχει πολλούς μηχανισμούς ασφαλείας και θα ήθελα να θέσω λοιπόν την εξής ερώτηση. Δεν θα πρέπει να σκεφτούμε πιο πολύ την ε, καλύτερη συνεργασία και ένα πιο σαφές σύστημα συνεργασίας μεταξύ των τριών αυτών ε, υπηρεσιών Ενδεχομένω δεν υπάρχει και άλλη υπηρεσία η οποία να εμπλέκεται στο πεδίο εφαρμογή αυτό. Ο κόσμο ε, προφανώ πλέον και περνάει από συστήματα πληροφορική και πληροφοριών, τα οποία και επισέρχονται σε όλου του τομεί τη καθημερινής ζωής πλέον. Όλα τα συστήματα λοιπόν αυτά συνήθως έχουν στρατηγική σημασία και θα πρέπει να τα προστατεύσουμε είναι ιδιαίτερως ε, ελκυστικά δε και για τους hackers, για οποιονδήποτε θέλει να κάνει επίθεση κατά αυτόν. Πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ των τριών αυτών ε, υπηρεσιών. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται οποιαδήποτε περίπλοκη νομοθετική ρύθμιση. Όχι. Νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε ποια θα είναι τα πιο δυνατά σημεία κάποια μεγάλα πλεονεκτήματα τη κάθε τέτοια υπηρεσία, προκειμένου τελικά ο κόσμο. να μην φοβάται ότι θα ανακύψουν προβλήματα σε περίπτωση επιθέσεων, για παράδειγμα, κατά των τραπεζών, στο ευρωπαϊκό σύστημα πλοήγησης. Αυτή είναι λοιπόν η ερώτηση που έχω να σας απευθύνω και θέλαμε να σα ευχηθώ και κάθε επιτυχία. Νομίζω ότι η θητεία σας είναι ιδιαίτερως δύσκολη γιατί Τώρα καλείστε να βρείτε καινούργιε στρατηγικέ και καινούργιε ιδέε για όλα αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σα. Μάλιστα. Έχουμε και εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων μαζί μας. Α, και ο οποίος δεν ήταν στον κατάλογο. Έχετε το λόγο. Κυρία Επίτροπε, ήταν πάρα πολύ ακριβή και αφήσει η παρουσίασή σας. Εγώ θα ήθελα να θέσω μία και μόνη ερώτηση σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξασφαλίσουμε. Αυτό όμως πώς μπορεί να το συνδέσουμε με την πτυχή της ασφάλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο. Και τώρα να ακούσουμε. Τελείωσαν οι πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ καταρχήν για τις ε, πολυάριθμες ερωτήσεις σας και την ενθάρρυνση που μου δώσατε γιατί ένα μεγάλο τμήμα ε, των ερωτήσεών σα αφορούσαν το πακέτο επιδεσμημέτρων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ευχαριστώ θερμά και το επιτελείο μου γιατί όλο το καλοκαίρι συνεχίσαμε τις προσπάθειες και την εργασία για το πακέτο αυτό για, το, για την κυβερνοασφάλεια. Να απαντήσω κατευχήν στον πρώτο ομιλήσατε, τον κύριο Μπόνι, για το χρονοδιάγραμμα και το ρυθμό του τριμερούς διαλόγου για τον κώδικα. Μάλιστα, η Κορεπέρ σήμερα συμφώνησε να προγραμματιστεί ο πρώτος τριμερής διάλογος για τις 25 Οκτωβρίου. Και μας εψυχώνει πολύ και μας εθαρρύνει ο δικός σας σταθερός ρυθμός. Το είπα και στην αρχή. Μας εθαρρύνει ιδιαίτερο στο γεγονός ότι η Επιτροπή Ήτρε κρατάει έναν αμύωτο ρυθμό στη διεκπαιρέωση των θεμάτων. Και αυτό μας εψυχώνει και εμάς και είναι κάτι που το είπα από την ανάληψη των καθηκόντων μου. Αν θέλουμε να υλοποιήσουμε την ενιαία ψηφιακή αγορά μέχρι τα τέλη του 2018, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Θα πρέπει τώρα να επιταχύνουμε το ρυθμό μας. Και επανέρχομαι αμέσως στο θέμα του φάσματος, γιατί όντως είναι ένα κρίσιμο ζήτημα και θα έλεγα, θα τολμούσα να πω ότι το φάσμα είναι ο άνθρακας και ο χάλιβα τη ψηφιακή οικονομία. και αυτό χρειαζόμαστε για να διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση. Και Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Έχουμε την εμπειρία και το κουράγιο των ιδρυτών πατέρων. Βέβαια, έχαμε πολλά ε, θαρρυντικά μηνύματα. Αλλά το πιο θεωρητικό ήταν ε, το, η διάσκεψη κορυφής του Τάλιν, η δέσμευση του Προέδρου Γιουνκέρ και τα θετικά μηνύματα που πήραμε από εκεί. Οπότε έχουμε ε, τη διάσκεψη κορυφής και 20 Οκτωβρίου, γιατί στη ψηφιακή διάσκεψη κορυφής του Τάλιν αναλύθηκαν κάποιες δεσμεύσεις άτυπα, θέλουμε να επισημοποιηθούν και επίσης έχουμε και το έκτακτο Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών. Και σίγουρα το φάσμα θα είναι από τα ε, κομβικά και νευραλγικά σημεία που θα εξεταστούν. Και όπως σας είπα, δεν θα αφιστώ προσπαθειών ώστε να συνειδητοποιήσουν τα κράτη-μέλη πόσο σημαντικά είναι αυτά τα θέματα γιατί αν χάσουμε σήμερα την ευκαιρία θα χάσουμε το τρένο. Μετά από 5-10 χρόνια θα είναι κατόπιν εορτής. Και το είδαμε και από ευκαιρία του 4G. Ε, χώρες που δεν ε, έχουν συντονιστεί και άλλες το εφαρμόσε σε 4 και άλλες 7 χρόνια δεν προχωράμε και θέλουμε να έχουμε πρωτοκαθεδρία στις νέες τεχνολογίες στο 5G, θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα στα θέματα αυτά και το μήνυμα μου θα είναι απερίφραστο προς όλα τα κράτη-μέλη. Όπου και αν πηγαίνω είναι από τα πρώτα θέματα που επισημαίνω. Σε ό,τι αφορά το κυβερνοπακέτο, καταρχήν, σε ό,τι αφορά την εντολή ε, του Οργανισμού για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών, του ΕΝΙΣΑ. Τέσσερα είναι τα πρωταρχικά στοιχεία. Καταρχήν, στην πρότασή μας έχουμε ε, την εντολή του ΕΝΙΣΑ που δεν είναι πια προσωρινή αλλά μόνιμη. Και αυτό έχει συγκεκριμένε συνέπειες. Πρόκειται για ένα σαφές μήνυμα σταθερότητας για τον οργανισμό, για το προσωπικό, αλλά και ένα μήνυμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση μακρόπνοης ε, προσέγγισης. Επίσης, τα επιχειρησιακά καθήκοντα της, ε, του ΕΝΙΣΑ προϋποθέτουν και ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Γι' αυτό και αυξήσαμε το προσωπικό του ΕΝΙΣΑ. Θα είναι 41 και ε, ο προϋπολογισμός θα περάσει από τα 11 στα 23 εκατομμύρια με 5 εκατομμύρια την πρώτη χρονιά λειτουργίας. Οπότε προτείνουμε ο οργανισμός ΕΝΙΣΑ να αναλάβει περισσότερα επιχειρησιακά καθήκοντα και μετά τις δημόσιες διαβουλεύσεις που είχαμε στις αρχές του έτους αναφέρει με σαφήνεια ότι ο Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών έχει την εμπειρογνωμοσύνη, έχει την τεχνογνωσία Οπότε θα πρέπει τώρα να αναλάβει το συντονιστικό του ρόλο μεταξύ των κρατών μελών, γιατί γνωρίζει την κατάσταση στα κράτη-μέλη, ε, οπότε μπορεί να δώσει ε, επιπλέον και μία όθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ε, μην ξεχνάτε και την οδηγία νης που είναι πολύ σημαντική και που λέει ότι η ενίσα είναι η γραμματεία, εξασφαλίζει το συντονισμό και είναι σημαντικό να μην παραμείνει σε γραμματιακό επίπεδο μόνο ο ΕΝΙΣ, ο οργανισμός ΕΝΙΣΑ. Γι' αυτό και δώσαμε πρωταρχικό ρόλο στον ΕΝΙΣΑ ό,τι αφορά την πιστοποίηση. Και έχετε δίκιο. Το σύστημα πιστοποίησης που προτείνουμε είναι προαιρετικό. Έχουμε θεωρήσει ότι δεδομένη στις πολυμορφίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δύο είναι οι βασικοί μας στόχοι. Καταρχήν, ένα περίφραστο μήνυμα προς το καταναλωτή και το χρήστη για να είναι σίγουρος για την ασφάλεια των προϊόντων και επίσης θέλουμε να επιτρέψουμε σε μια εταιρεία που έχει πιστοποιητικό σε ένα κρατός μέλος να αναγνωρίζεται και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις γιατί μειώνει το κόστος και την επιβάρηση. Ξέρετε τι τιμή έχουν τα πιστοποιητικά από τη μια χώρα στην άλλη η ψαλίδα είναι από 150.000 μέχρι 300.000 ευρώ. Μεγάλη διαφορά. Επίσης, ε, οι κρίσιμες ε, υποδομές σε κάποιους τομείς είναι πολύ σημαντικές. Ε, οπότε, διερευνούμε και την πιθανότητα η πιστοποίηση αυτή να γίνει υποχρεωτική για κάποιους τομείς. Αλλά ας αφήσουμε τον ίδιο τον κλάδο που έχει την εμπειρογνωμοσύνη μαζί με τον Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών να ε, δει ποια θα είναι η ακολουθητέα απόρία. Σε ό,τι αφορά το σύστημα προειδοποίησης. Αυτό το σύστημα συνδυάζει δύο τεινά. Καταρχήν, για πρώτη φορά σε πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέσαμε σε αυτό το blueprint που λέμε τη στρατηγική. Αυτό έχει απήχηση στους Ευρωπαίους πολίτες, γιατί τι σημαίνει Ευρωπαϊκός Μηχανισμός ε, Συντονισμού σε περίπτωση επιθέσεων μεγάλης κλίμακος, Σήμερα δεν γνωρίζουμε ποιο είναι αρμόδιος γιατί. Και είχαμε χαρακτηριστικά παραδείγματα και χάρη στην πρότασή μας υπάρχει αυτή η δυνατότητα πια συντονισμού. Σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, τον κλάδο και τα θεσμικά όργανα προτείνουμε ένα πλαίσιο συντονισμού σε περίπτωση επιθέσεων μεγάλης εμβέλειας. Επιπλέον, ο ΕΝΙΣΑ που μέχρι στιγμής ε, ε, κάθε δύο χρόνια... Ε, ε, είχε κάνει αξιολόγηση για να δει τις αδυναμίες των κρατών μελών. Τώρα θα γίνεται ετησίω αυτή η αξιολόγηση. Και το blueprint θα ελεγχθεί για πρώτη φορά στην επόμε, την επόμενη φορά. Επίσης, όταν μιλούμε για σύστημα προειδοποίησης, ε, το θέμα του ΣΕΡΤ είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια κεντρική μονάδα που έχει τους ομολόγους και τους συνομιλητές στα κράτη-μέλη. Θέλουμε αυτό το κέντρο να είναι διαθέσιμο συνέχεια, 24 ώρες 24 ώρες, 7 μέρες τη βδομάδα. Είναι σημαντικό λοιπόν και στην οδηγία έχουμε τη δυνατότητα επιχειρησιακών δραστη... Ε, ικανοτήτων για το ΕΝΙΣΑ, για το κέντρο αυτό, ώστε να αναβαθμίσουμε το επίπεδο κυβερνοασφάλειας, κάτι που επιθυμούμε όλοι. Και στον κανονισμό για τον ε, ΕΝΙΣΑ θα έχουμε την πρόταση για το ΣΕΡΤ, ε, για την Επιτροπή Ενέργειας Έρευνα και Τεχνολογίας και θέλουμε μία μονάδα που να εκπροσωπεί το, συγγνώμη, την ομάδα παρέμβαση για συμβάντα που αφορούν την ασφάλεια των υπολογιστών. Υπάρχει μία μονάδα στις Βρυξέλλες που μπορεί να ανταποκρίνεται με τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Πρόκειται για συγκεκριμένες προτάσεις, συντονισμός δηλαδή, ταυτόχρονα σύστημα πιστοποίηση, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα για τον κλάδο, τους καταναλωτέ και για, τους, ε, τον υπόλοιπο κόσμο. Και επίσης ε, λέμε ξεκάθαρα ότι ε, τη σήμερον ημέρα δεν μπορεί ένα κράτος μέλο μόνο του να αντιμετωπίσει μία κυβερνοεπίθεση. Θα πρέπει να συντονιστούμε και να συνεργαστούμε. Αυτά για τις πρώτες ερωτήσεις. Τώρα κύριε Τοσενόφσκι για τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των τριών οργανισμών. Ε, ένα ζήτημα πολύ ευαίσθητο. Πήγα στο οργανισμό ΕΝΙΣΑ πριν από λίγες εβδομάδες στην Ελλάδα και είχα συζήτηση με το προσωπικό. Ρώτησα λοιπόν, πόσο συχνά ανταλλάσσετε πληροφορίες ε, με τους υπόλοιπους οργανισμούς. Ποτέ, μου λένε. Θα πρέπει λοιπόν να εγγύψουμε και σε αυτό το σημείο σήμερα, το συντονισμού των οργανισμών, για να δούμε με ποιου μηχανισμού μπορούμε να εξασφαλίσουμε τέτοιο συντονισμό. Πολλά δε μάλλον που έχουμε μια ειδική, ε, ειδική υπηρεσία, ένα ειδικό οργανισμό για την ασφάλεια, την κυβερνοασφάλεια. Οπότε θα πρέπει η ανταλλαγή πληροφοριών να γίνεται, όχι απαραίτητα με υλική παρουσία, σωματική παρουσία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να το παραβλέπουμε γιατί σήμερα οι κυβερνοεπιθέσεις δεν μας θίγουν προσωπικά ή σε θεσμικό επίπεδο μπορεί να έχουν εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες ακόμη και στο σύστημα υγείας, στα ενεργειακά συστήματα, στα συστήματα μεταφορών. Είναι πραγματικά μια τεράστια πρόκληση. Και κύριε Νίκα για την επιχείρηση Κασπέρσκι που αναφέρατε. Δεν είμαι μόνη αρμόδια για το θέμα αυτό, αλλά θα επανέλθω στο θέμα αυτό και θα επισημάνω το πρόβλημα στην κυρία Φερστάγκερ, γιατί είναι θέμα και ανταγωνισμού. Πάντως συνεργαζόμαστε πολύ καλά με την Επίτροπο Φερστάγκερ, έχουμε τακτικές επαφές, οπότε θα της αναφέρω το ζήτημα και θα σας ενημερώσω μόλις συγκεντρώσω τις απαραίτητες πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ακούσουμε τώρα τους άλλους ομιλητές. Βέρνερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ και καλώ ορίσατε και από δική μου πλευρά, αγαπητή κυρία Επιτροπή. Θα ήθελα να σα κάνω κάποιε ερωτήσει για το πακέτο τη ε, ασφάλειας. Γιατί πολλέ μικρομεσαίε επιχειρήσει ε, φοβούνται την περαιτέρω ψηφιοποίηση ακριβώ γιατί έχουν ανησυχίε για την ασφάλεια των δεδομένων τους και δεν είναι και δικαιολόγητη αυτή η ανησυχία γιατί η κυβερνοασφάλεια και οι επιθέσεις σε αυτή έχουν ε, πολύ μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις και μάλιστα αυτές επιταχύνονται και έχουν πενταπλασιαστεί τελευταία χρόνια. Με ακούτε, με ακούτε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό κάποιο πρόβλημα φαίνεται να υπάρχει. Στην τα ακουστικά της Επιτρόπου. Συγγνώμη, συγγνώμη λέει ο Πρόεδρος, γιατί Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. It's working. Try, try once, once again. Θέλετε να ξαναξεκινήσετε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα ξεκινήσω λοιπόν από την αρχή. Θα ήθελα λοιπόν να σα κάνω κάποιε ερωτήσει σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Καλώ ορίζω καταρχά το γεγονό, το πακέτο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό γιατί πολλέ μικρομεσαίε επιχειρήσει ε, ανησυχούν και δεν προτιμούν την περαιτέρω ψηφιοποίηση γιατί ανησυχούν για την ασφάλεια των δεδομένων του. Και αυτό δεν είναι δικαιολόγητο γιατί οι οικονομικέ επιπτώσει ε, των κυβερνοεπιθέσεων έχουν πενταπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Και έτσι λοιπόν με την διασύνδεση αυτή η τάση θα συνεχίσει να αυξάνεται. Βρισκόμαστε λοιπόν στην εξή κατάσταση. Έχουμε όλο και πιο πολλέ ε, μικρομεσαίε επιχειρήσει που πλήττονται από τι κυβερνοεπιθέσει και συχνά με ναι, καταλαβαίνετε, πολύ ωραία. Και συχνά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο στον οποίο διατρέχουν. Δεν έχουν άλλωστε και τους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη προκειμένου να εφαρμόσουν μια αυστηρή πολιτική ασφάλεια στην επιχειρήση. Και Πώ υποστηρίζονται λοιπόν αυτέ οι επιχειρήσει με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ασφάλεια. πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων και τα κενά στην ασφάλεια. Συχνά ακούμε για τα προβλήματα του λογισμικού. Το security λοιπόν η ασφάλεια ε, κατά το σχεδιασμό δεν είναι κάτι το οποίο είναι ευρέως δεδομένο. Πώς μπορείτε επίσης ε, να διευρύνεται το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία για την ασφάλεια για να περιλαμβάνει και το λόγο γενικό. Τελευταία ερώτηση. Το Μάιο του 2017 οι κυβερνοεπιθέσει και η μεγάλη αύξηση τέτοιων ε, περιπτώσεων απάτη ε, ε, για το fake residency ουσιαστικά κατέδειξαν ότι λείπουν βασικές ικανότητες ψηφιακής, αν θέλετε, ικανότητας ε, στον κόσμο, στους πολίτες. Και μιλάμε για έναν τέτοιο κλάδο ο οποίος αυξάνεται όλο και πιο πολύ. Πώς λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το πακέτο που προτείνει μπορεί να βοηθήσει προκειμένου να υπάρχει καλύτερη αντίληψη και συνειδητοποίηση των κινδύνων αυτών που τρέχει και των μέσων προστασία που μπορεί να λάβει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρο. Η κυρία Νίμπλερ είναι η επόμενη ομιλητρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα από πλευρά μου να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω την Επίτροπο. Σα ευχαριστώ για τον δυναμισμό τον οποίο ε, καταδεικνύεται στα νέα σα καθήκοντα και νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ φιλόδοξο το πρόγραμμα το οποίο έχετε. Οι συνάδελφοι έδειξαν το θέμα της κυβερνοασφάλεια και εγώ θα ήθελα λοιπόν να σα συγχαρώ για την πρόταση την οποία καταθέσατε. Πιστεύω ότι είναι καλό το ότι διευρύνεται το πεδίο εφαρμογή τη ΕΝΙΖΑ, προτείνεται και απόψει προσωπικού και από απόψει ε, πόρων να υπάρχει καλύτερο εξοπλισμό τη θενίζα και σε ό,τι αφορά τι εργασίε τη, θα πρέπει να συζητήσουμε λεπτομερέστερα το τι θα γίνει, αλλά η προσέγγιση είναι καλή. Έχω μια ερώτηση, Η πρώτη ερώτηση σε ό,τι αφορά αυτά τα μόλις, ε, που μόλι μα είπατε. Είπατε, κύριε Επιτροπέ, ότι σε ό,τι αφορά τις αθέμητες ε, εμπορικές πρακτικές των ε, πλατφόρμων online θέλετε να τις καταπολεμήσετε αυτές τις αθέμητες πρακτικές και θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε σε ποια κατεύθυνση σκέφτεστε να κινηθείτε. Στις πλατφόρμες θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά κατά περίπτωση. Αυτές οι πλατφόρμες που έχουν ε, τη λειτουργία τήρησης των δεδομένων θα πρέπει να δούμε τι δομές διαχείρισης μπορεί να προκύψουν. Δεύτερη ερώτηση που θέλω να σας θέσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε προτάσει νέων φορολογικών διατάξεων για τους tech giants, για τις μεγάλες αυτές επιχειρήσεις. Πείτε μας λίγο παραπάνω και γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο Δεν ονατώ. Α, όχι, συγγνώμη. Σωρίνιο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Επίτροπο να την συγχαρώ θερμά για τον πολύ επαγγελματικό τρόπο και τη μεγάλη εργατικότητα και επιμέλεια με την οποία προσέγγισε τα έτσι καθήκοντα. Ε, και, και χαίρομαι και για τη σημασία που δώσατε στην πρωτοβουλία Wi-Fi for Europe. Φάνηκε από τη συζήτηση ότι το κεντρικό ζήτημα που είναι η βάση των πάντων, είναι η οικονομία των δεδομένων, η σωστή χρηστή διαχείριση των δεδομένων, ώστε με τα δεδομένα να μεταβιβάσουμε ασφάλεια στους ε, Ευρωπαίους, να μεταδώσουμε ασφάλεια. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το κλειδί των πάντων είναι η ασφάλεια για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ασφάλεια απέναντι στην τρομοκρατία και το έγκλημα. Αλλά ασφάλεια απέναντι και στην επισφαλή απασχόληση. Ασφάλεια απέναντι στις κλιματικές αλλαγές, στις θεομηνίες και φυσικές καταστροφές, την ιδιωτική του σφαίρα, τα ατομικά τους δικαιώματα. Και όλα αυτά εξαρτώνται από τα δεδομένα, την σωστή διαχείριση και σωστή ανταλλαγή δεδομένων. Όλα αυτά εξαρτώνται από μία ευφύ ε, διαχείριση αυτού του τεράστιου πλούτου που έχουμε με τα δεδομένα. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε αυτή την επιθυμητή ασφάλεια, χωρίς όμως να θυσιάσουμε την ιδιωτικότητα. Και να δούμε πώς, τι επικοινωνιακό τρόπο θα διαλέξουμε για να μην μεταδώσουμε φόβο αντί για ασφάλεια ή να μην ε, επιδεινώσουμε την ανησυχία του κόσμου ή να μην επιβαρύνουμε υπερβολικά τι επιχειρήσει. Δηλαδή, ανταλλαγή δεδομένων για να αποτρέψουμε την τρομοκρατία και το έγκλημα, για να βελτιώσουμε την επιχειρηματικότητα, να δημιουργήσουμε νέε θέσει απασχόληση, να φέρουμε τη διοίκηση τη δημόσια διοίκηση πολύ πιο κοντά στους πολίτες, ιδιαίτερα όταν είναι συρρυκνωμένοι οι κρατικοί προϋπολογισμοί. Επίσης, δεδομένα για τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Έρευνας και κοινοτομία, για να γίνουν πιο ανταγωνιστικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Κύριε Επίτροπε, είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε αυτό το πλαίσιο εμπιστοσύνη και να θέσουμε τα δεδομένα στην υπηρεσία των, της ασφάλειας, χωρίς να διαταράξουμε όμως ή να διαρρήξουμε την ιδιωτική σφαίρα. Συγχαρητήρια πραγματικά για το έργο σας. Μπορείτε λοιπόν να ξεκινήσετε μια εκστρατεία επικοινωνίας για να μεταδώσουμε σωστά όλα αυτά τα θέματα στους Ευρωπαίους πολίτες. Σας ευχαριστώ κύριος Κρασνοντέμψκι. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπό για την ελεύθερη ροή των μη προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγματικά αυτό είναι πολύ σημαντικό το βήμα της πρότασής σας και στην πατρίδα μου ήμασταν υπέρμαχοι ε, υπέρ της πρωτοβουλίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να καταργηθούν αυτά τα αδικαιολόγητα προσκόμματα σε αυτήν την ελεύθερη ροή των μη προσωπικών δεδομένων. Φαίνεται όμως ότι δημιουργείται μια ατμόσφαιρα αυξανόμενου προστατευτισμού. Θα συζητήσουμε και την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων. Διαπιστώνουμε ότι όλο και περισσότερο αφισβητείται το θέμα αυτό. Ε, και μιλούμε για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Για, από τη στιγμή που θέλουμε ενιαία ψηφιακή αγορά θα πρέπει να καταργήσουμε τα περιτά και τα δικαιολόγητα εμπόδια. Ε, μια άλλη ερώτηση αφορά την ασφάλεια. Γιατί εξαίρεση θα είναι τα δεδομένα που θα αφορούν θέματα εθνικής ασφάλειας. Ποια κριτήρια θα υιοθετήσει, σπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να περιορίσει τα δεδομένα και πώς θα κρίνει τέτοιου είδους δραστηριότητες. Άλλη ερώτηση. Το θέμα της συνεργασίας με τα σημεία επαφής που θα εγκατασταθούν στα κράτη-μέλη και που θα υλοποιήσουν, θα εφαρμόσουν τον κανονισμό. Και αυτό θα είναι κέριο σημείο. Πώς θα συνεργάζονται μεταξύ τους τα σημεία επαφής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να ρυθμίσει αυτό το συντονισμό και αυτή τη συνεργασία στο μέλλον μήπως θα θεσπίσει το μέλλον και εφαρμοστικές εκτελεστικές πράξεις ως προς αυτό. Επίσης, ε, κώδικα συμπεριφοράς ε, για τους επιχειρηματίες. Καλό θα είναι αυτό να γίνει ε, κάτωθεν, από τη βάση δηλαδή, και δεν ξέρω με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να στηρίξει αυτές τις αυτορυθμιστικές προσπάθειες. Σας ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις σας. Κύριε Επίτροπε, από ό,τι βλέπω δεν ζητά άλλος κανείς συνάδελφος το λόγο για να υποβάλει ερωτήσεις, οπότε αυτός είναι και ο τελευταίος γύρος των απαντήσεών σας. Και μπορείτε να κάνετε και την ανακεφαλαίωση στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Όσον αφορά τις μικρομισές επιχειρήσεις καταρχάς. Όντως, ε, ως Επίτροπος, δεν πρόκειται να παραβλέψω προφανώς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προφανώς θα πρέπει, δύο σημερινή εποχή, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε βέλτιστες πρακτικές, να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών. Ένα 80% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων λένε ότι έχουν ε, πέσει θύμα κυβερνοεπίθεσης μέσα στο τρέχον αυτό έτος. Και άλλες επιχειρήσεις μας λένε ότι κάθε φορά που μιλάμε για κυβερνοεπιθέσεις υπάρχουν δύο ομάδες προσώπων, αυτοί που γνωρίζουν ότι ήταν θύματα επίθεσης και αυτοί που ακόμα το αγνοούν. Σας ευχαριστώ πολύ που θέσετε λοιπόν το ζήτημα αυτό. Στο σημερινό κόσμο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να μιλήσουμε όλο και περισσότερο για αυτό το οποίο αποκαλούμε κυβερνοϊγιεινή, πρακτικές αντιμετώπισης των κυβερνοεπιθέσεων, καθότι ε, ξέρετε ότι ε, πάρα πολλές επιθέσεις συνδέονται και με τη γενικότερη αυτή τάση παραπληροφόρησης και πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ήδη πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα αυτά. Ήδη τώρα από το μήνα Οκτώβριο έχουμε αρχίσει να επιμένουμε περισσότερο στο ζήτημα της κυβερνοασφάλειας και ξέρετε ότι ήδη από τον μήνα Οκτώβριο στις εκδηλώσεις που έχουμε ήδη οργανώσει έχουμε προσκαλέσει πολλές ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα θέλαμε και στο μέλλον να έχουν πρόσβαση στις διαβουλεύσεις που λαμβάνουν χώρα. Και Κάτι ακόμα. Είπα ότι ενδεχομένως θα δημιουργήσουμε κέντρα έρευνας και δεξιοτήτων σε διάφορα κράτη-μέλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι εμπειρογνώμονε, οι οποίοι ήδη γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα για τα ζητήματα αυτά τη κυβερνοασφάλεια, να μπορούν να διοχετεύσουν τη γνώση του αυτή. Είναι σημαντικό να μπορούμε να έχουμε ακόμα και καταρτήσει στα τη κυβερνοασφάλεια αυτά τα κέντρα δεξιοτήτων και έρευνα. Και έπειτα και την στρατηγική για την ψηφιοποίηση τη βιομηχανία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κόμβους ψηφιακής καινοτομίας. Έχουμε ήδη προπολογισμό για τα επόμενα τρία χρόνια, 300 εκατομμύρια ευρώ, και επομένως θα πρέπει να συμπεριλάβουμε ακόμα και την, την πτυχή αυτή σε, αυτά στις, σε αυτούς τους κόμβους ψηφιακής καινοτομίας. Ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πολλές φορές δεν καταφέρνουν λόγω της γεωγραφικής τους θέσης να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, να μπορούν να συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά. Κυρία Νίμπλερ, ξέρετε ότι σε σχέση με την παρατήρηση που κάνατε με τον Επίτροπο Μοσκοβισή και με την Επίτροπο Βεστάγκερ, ασχοληθήκαμε με το ζήτημα αυτό και προχωρήσαμε μάλιστα και σε μια ανακοίνωση. Είπαμε ότι μέχρι το Δεκέμβριο, μαζί με τους εταίρους μας από τον ΩΣΑ, θα προωθήσουμε την πρόταση αυτή, αλλά αν δεν ευοδοθεί τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει μόνη της. Ξέρετε λοιπόν ότι έχουμε ήδη ένα συγκεκριμένο στόχο και δεν ε, τον χάνουμε αυτόν από τον ορίζοντα. Θέσατε επίσης και ένα ερώτημα, ερώτημα με συγχωρείτε, που έχει να κάνει με τις αθέμητες ε, πρακτικές. Ξέρετε ότι και με το ζήτημα αυτό θέλω να ασχοληθώ. Ήδη από τις αρχές του 2018 θα υποβάλω μια νομοθετική πρόταση όσον αφορά τις ε, αθέμητες πρακτικές. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάθε φορά να μπορούμε να προωθούμε την δική μας προσέγγιση θα επεμβαίνουμε κάθε φορά που θεωρούμε ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία ή θα επεμβαίνουμε εκεί πέρα στους τομείς εκείνους που θεωρούμε ότι θα πρέπει να, να προστατευτούν περισσότερο τα δικαιώματα των καταναλωτών. Σαφώς συνειδητοποιούμε ότι οι πλατφόρμες αποτελούν κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη, αλλά παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα σε δικαιοσύνη, αξίες και κοινοτομία και πιστεύω ακράδαντα ότι εκεί έγκυται πραγματικά η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι μπορούμε μέσω των τριών αυτών πτυχών που έθιξα να ε, καθορίσουμε συγκεκριμένου κανόνες. Κύριε Ζωρίνιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το Wi-Fi for EU, το project αυτό, το σχέδιο αυτό μας ενδιαφέρει όλους ιδιαιτέρως. Θα ολοκληρώσουμε την σχετική διαδικτυακή πύλη μέχρι το τέλος του έτους και τα πρώτα κουπόνια θα ε, γίνουν διαθέσιμα ήδη από τις αρχές του 2018. Σας το είχα πει αυτό και στην συζήτηση που κάνουμε κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας, αλλά θα επανέλθω στο ζήτημα αυτό. Κάθε φορά που μιλάμε για ανταλλαγή δεδομένων, τίθεται πάντα το ζήτημα της εμπιστοσύνης των πολιτών. Αυτό έχει θεμελιώδη σημασία. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε μια ενημερωτική εκστρατεία προκειμένου να ενημερώσουμε τους πολίτες για όλα αυτά τα μέτρα τα οποία υιοθετούμε. Όσον αφορά τώρα την ελεύθερη κυκλοφορία των μη προσωπικών δεδομένων, κύριε Κρασνοντεύσκη, όντω, η Πολωνία βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της πρωτοβουλίας αυτής. Ήδη χθε το βράδυ ήμουνα μαζί με τον Κριστόφ Σουμπέρα σε μια τέτοια εκδήλωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι η οικονομία των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχεί σε 257 δισεκατομμύρια ευρώ, 2% του ΑΕΠ και θέλουμε να φτάσουμε στο 4% του ΑΕΠ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο υποβάλαμε την πρόταση αυτή για την ελεύθερη ροή των μη προσωπικών δεδομένων. Κάθε φορά όμως αυτό, το κάνουμε αυτό θα πρέπει να γίνεται ε, με απόλυτο συντονισμό των διατάξεων που προβλέπονται στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων, του GDPR. Στην πρότασή μας λοιπόν, μόλον ότι θα προωθήσουμε προφανώς την ροή των δεδομένων αυτό, θα πρέπει να τηρούνται και οι διατάξεις του Γενικού Αυτού Κανονισμού. Όσον αφορά τώρα τη συνεργασία μεταξύ των σημείων επαφής επί του παρόντος, δεν προχωρήσαμε καθόλου σε εκτελεστικές ή άλλες νομοθετικές αποφάσεις. Όπως και στην περίπτωση των πιστοποιήσεων, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε σε μια πρώτη φάση πώς λειτουργεί στην πράξη το σύστημα αυτό. Η οδηγία νης για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών δεν έχει ακόμα αρχίσει να εφαρμόζεται. Επίσης θέλουμε να προχωρήσουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα με την ε, κυβερνοασφάλεια και τη ροή των μη προσωπικών δεδομένων, όσο πιο γρήγορα αρχίσουν να εφαρμόζονται οι προτάσεις αυτές στην πράξη, τόσο πιο γρήγορα θα καταφέρουμε να δούμε αν τελικά συνεργάζονται αποτελεσματικά τα σημεία επαφή και εν συνεχεία θα είμαστε σε θέση να κάνουμε μια πιο ενδελεχή ανάλυση για τη μεταξύ των σημείων αυτών συνεργασία και για το αν θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω βελτιώσει. Αυτά είχα να σα πω. Ελπίζω να απάντησα στι παρατηρήσει και τι ερωτήσει σα. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτόν τον πρώτο διαρθρωτικό διάλογο που έχω σήμερα εδώ μαζί σα. Διατηρώ, όπω πάντα, τον αρχικό μου ενθουσιασμό και χαίρομαι πάρα πολύ που για άλλη μια φορά με δεχτήκατε τόσο θερμά στην Επιτροπή σας. Επαναλαμβάνω τη βούλησή μου να συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί σας με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και όσο το δυνατόν πιο επικοδομητικά γίνεται. Μαζί θα δημιουργήσουμε την ψηφιακή ενιαία αγορά και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που προασπίζει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προτάσεις αυτές οι οποίες εμπλουτίζουν το νομοθετικό μας έργο και που αντικατοπτρίζονται τελικά στην τελική εκδοχή των νομοθετικών μας αποφάσεων. Ξέρετε ότι μέσω της συνεργασίας αυτής θα πρέπει πραγματικά να εξυπηρετηθούν οι πολίτες μας. Αυτοί βρίσκονται στο κέντρο των αποφάσεών μας και πιστεύω ότι πάρα πολλές προκλήσεις θα καταφέρουμε να τις αντιμετωπίσουμε στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας. Μάλιστα. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν τη συζήτησή μα, ήταν πάρα πολύ καλέ αυτά τα σχόλιά σα, αλλά μήπω κάποιοι συνάδελφοι ήθελαν να πάρουν το λόγο, γιατί νομίζω ότι έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο, αν μου επιτρέπετε. Ήταν πραγματικά πολύ καλή η εισήγησή σα. Ευχαριστώ κύριε Σουσαν Κέλλη, ευχαριστώ πρόεδρε και συγγνώμη που καθυστέρησα γιατί ήμουν στο Ευρωπαϊκό Βραβείο για τους πολίτες, του πολίτη. Χαιρόμαστε που είσαστε εδώ πέρα λοιπόν μαζί μα. Κάποιες ερωτήσεις να σας κάνω για την κυβερνοεπίθεση το Μάιο του 2017. Μας υπενθυμίζει την, ε, τους κινδύνους που υπάρχουν στις πολίτες σε ένα όλο και πιο ψηφιωμένο κόσμο. Και θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια απάντηση για την ασφάλεια για να έχουμε μεγαλύτερη ικανότητα προστασία του πολίτη από τέτοια περιστατικά. Αλλά να επιστήσω την προσοχή σα στο εξή. Μια έκκληση τη Microsoft και άλλων επιχειρήσεων για μια, για μια ψηφιακή σύμβαση τη Γενέβη, ε, τη Γενέβη. Ε, υπάρχει ένα αιτήσιο συνέδριο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα σε παγκόσμιο επίπεδο γιατί είναι παγκόσμιο ζήτημα. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν, σχολιάστε. Πιστεύετε ότι θα υπήρχε μια τέτοια δυνατότητα χωρίς να μπείτε σε μεγάλο βαθμό λεπτομέρειες και σας ευχαριστώ πρόεδρε που μου επιτρέψατε να κάνω την ερώτηση αυτή. Μάλιστα, από ό,τι βλέπετε, ήταν καλή η τελευταία αυτή ερώτηση. Ε, πρόκειται για ένα παγκόσμιο ζήτημα αυτή τη φορά. Κοιτάξτε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη και πολύ συγκεκριμένη μάλιστα και το επόμενο ραντεβού θα είναι στη Γενέβη στις 18 μέχρι 22 Δεκεμβρίου και ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πάντα καλά εκπροσωπούμενο ε, και σε ό,τι αφορά τις παγκόσμιες ε, προκλήσεις και την κυβερνή ασφάλεια και εγώ έχω ήδη επιβεβαιώσει ότι θα παραστώ στο συνεδρίο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέει ο Πρόεδρος. Ε, Επίτροπε, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισκέψή σας στην Επιτροπή Ήτρε και από ό,τι βλέπετε μας ε, ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα ψηφιακά ζητήματα. Έχουμε λοιπόν ε, την ψηφιακή ένωση κατάνω, Δεν μας φτάνει η ψηφιακή ενιαία αγορά. Ενδεχομένω να μην είμαστε έτοιμοι να τα όλα αυτά στην τρέχουσα θητεία, αλλά Προετοιμαζόμαστε για την επόμενη, τα επόμενα πέντε χρόνια και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα πούμε βεβαίως ε, συντόμως, ελπίζουμε. Ευχαριστώ. Uh, Και κυρίες και κύριοι θα συνεχίσουμε Πάρα αυτά στο επόμενο ζήτημα της ημερήσιας δέταξης. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν θα ήθελα να σας διαβιβάσω ένα σύντομο μήνυμα ενημερωτικό. Σήμερα το απόγευμα θα έχουμε μαζί μας δύο ομάδες ε, επισκεπτών στην συνεδρίαση. Μία ομάδα 15 δημοσιογράφων από τη Δανία, καλεσμένοι του κυρίου Πέτερσεν, που καλύπτουν ε, και τρέχουν ε, θέματα ενεργείας, καθώς και μια ομάδα επισκεπτών της κυρίας Βέρνερ, η οποία θα καταφτάσει αργότερα. Καλωσορίζουμε λοιπόν τα μέλη των δύο αυτών ομάδων επισκεπτών στην ε, Επιτροπή μας και πρώτα απ' όλα την ομάδα του κυρίου Πέτερσεν. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Και τώρα να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. διαπραγματευτική εντολή για τον αγωγό Nord Stream 2 κατάσταση των πραγμάτων παρουσίαση από τον Klaus Dieter Borchardt, διευθυντή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Γενική Διεύθυνση Ενέργειας προφανώς. Όπως τα ξέρετε δε και θα θυμάστε, στις 12 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μία σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της έναρξης διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη λειτουργία του αγωγού Nord Stream 2. Θα γνωρίζετε ότι εμείς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχαμε την ευκαιρία να δούμε και να εξετάσουμε με ιδιαίτερο τρόπο αυτή την πραγματική εντολή. Σήμερα λοιπόν πολύ σημαντική η συνάντησή μα. Ο, Κλάους, ο κύριος Κλάου Δίτερ Μπορχάρτ, διευθυντή τη Γενική Διεύθυνση Ενέργεια, θα ενημερώσει την Επιτροπή μα, την Επιτροπή Ήτρα, για τι τελευταίε εξελίξει σε ό,τι αφορά τα σημαντικά αυτά ζητήματα, το σημαντικό αυτό φάκελο και για τι συζητήσει στο Συμβούλιο. Να προσθέσω δε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι η επόμενη ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για το Nord Stream 2 προγραμματίζεται για αύριο. Αύριο 12 Οκτωβρίου. Άρα η συζήτησή μας ε, έρχεται σε κέριο χρονικό σημείο. Κύριε Δευθυντά, έχετε το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ καθηγητέ Μπούζεκ, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, μέλη της Επιτροπής Ήτρε, με μεγάλη χαρά θα σε ενημερώσω σήμερα για την κατάσταση των συζητήσεων σε ό,τι αφορά την εντολή για τον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2. Πριν ε, σας ενημερώσω όμως ε, για το πώς έχουν τα πράγματα, θα ήθελα να επισημάνω και να επαναλάβω την προσήλωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής του στόχους της Ενεργειακής Ένωσης και κυρίως την εξασφάλιση της του, της ενεργειακής ασφάλειας και στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Προτεραιότητά μας είναι να έχουμε μια ανταγωνιστική και διαφοροποιημένη αγορά φυσικού αερίου. Είναι σαφές επίσης ότι το σχέδιο ε, φυσικού αερίου, αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2 υπονομεύει την προτεραιότητα που σας προανέφερα. Και να σας ε, πω με δύο λόγια το σκεπτικό μας. Δεδομένου του μεγέθους των διαστάσεων, γιατί μιλάμε ε, για 55 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο. Για έναν αγωγό δηλαδή που θα επηρεάσει αισθητά τη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς και την ασφάλεια του ανεφοδιασμού. Ε, και αντιβαίνει στις προσπάθειες διαφοροποίησης ε, ε, πολλών κέντρων ανατολικών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης σε μεγάλο βαθμό παρακάμπτει την διαμετακόμιση φυσικού αερίου, τη διέλευση φυσικού αερίου από την Ουκρανία. Πώς καταλήξαμε σε αυτό το συμπέρασμα. Αν σκεφτείτε ότι ένα μόνο μέρος συμβαλόμενο, η Gazprom, έχει περιορίσει την πρόσβαση στην μεγαλύτερη αγορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη, τη Γερμανία δηλαδή, αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των αγορών και το διασυνοριακό εμπόριο με τις γειτονικές χώρες. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του ανεφοδιασμού, θεωρούμε ότι ο αγωγός Nord Stream 2, ακριβώς επειδή θα συγκεντρώνει τεράστια δυνατότητα μεταφοράς, δηλαδή 55 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα από το Nord Stream 2, και σε αυτό θα πρέπει να προσθεθεί γιατί περνάει από το ίδιο βόρειο διάδρομο του Nord Stream 1 που επίση έχει άλλα 55 δισεκατομμύρια. Δηλαδή μιλούμε για 110 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα που θα περνάνε από το βόρειο διάδρομο. Αυτή λοιπόν η υπερβολική συγκέντρωση σε ένα σχετικά μικρό διάδρομο όπως είναι ο Βόρειος, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οποιαδήποτε διαταραχή στο διάδρομο αυτό θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος και άρα και την ασφάλεια του ανεφοδιασμού. Πάνω από το 80% του συνόλου των ρωσικών εξαγωγών θα περνάνε μέσα από αυτό τον ένα και μόνο διάδρομο. Και η διοχέτευση τόσο μεγάλων ποσοτήτων φυσικού αερίου από ένα και μόνο διάδρομο, το Nord Stream, θα αποβεί βάρος όπως σας εξήγησα και του ουκρανικού, της ουκρανικής διαμετακόμισης, γιατί εμείς δεν πιστεύουμε όπως λένε οι Ρώσοι, όπως ε, θέλω να πιστεύουμε μερικά κράτη-μέλη, ότι αυτά τα 55 δισεκατομμύρια είναι επιπλέον ποσο, ποσότητες. Κατά τη γνώμη μας είναι αναδιοχέτευση, δεν είναι συμπληρωματικές ποσότητες. Παρακάμπτεται απλώς η Ουκρανία. Και η Ρωσία πολλές φορές δήλωσε ότι θέλει να περιορίσει τις ποσότητες αυτές από τη διαμετακόμιση, από τη διέλευση τους από την Ουκρανία. Κάτι τέτοιο επίσης σημαίνει ότι οι νότιο-ανατολικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επηρεαστούν, γιατί ε, τώρα αυτό το αέριο θα πηγαίνει στους δυτικούς κόμβους. Αλλά άρα η νότιο-ανατολική Ευρώπη θα πρέπει να εφοδιάζεται από τη Δύση, δηλαδή μεταφορά σε μεγαλύτερες αποστάσεις και άρα ε, υψηλότερε τιμέ για την Νότια Ανατολική Ευρώπη και χώρε που ήδη αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα θα πρέπει να πληρώνουν υψηλότερε τιμέ φυσικού αερίου. Ενώ οι δυτικέ αγορέ θα έχουν και πολύ προσιτέ τιμέ, καλέ τιμέ και καλύτερη εξυπηρέτηση. Ενώ οι νοτιοανατολικέ χώρε θα πληρώνουν ε, υψηλότερο κόστος μεταφοράς και σε τελική ανάλυση ακριβότερο φυσικό αέριο. Δεδομένου λοιπόν όλων αυτών των συνεπειών και αυτού του αντικτύπου, Θεωρώ ότι θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ σημαντικό αυτός ο αγωγός φυσικού αερίου να ε, περιορίζεται από ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο. Ποιο είναι αυτό όμως το σαφές κανονιστικό πλαίσιο. Η νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρόσφατα και η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου έκριναν ότι η οδηγία για το φυσικό αέριο δεν εφαρμόζεται άμεσα σε εξωχώριους φυσικούς αγωγούς όπως θα είναι ο Nord Stream που θα είναι υποθαλάσσιος εντάξει θα έλεγα. Έχει καλός. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα αφήσουμε αυτό τον αγωγό σε ένα νομικό κενό ή ακόμη χειρότερα θα αποδεχθούμε ότι ο αγωγός αυτός ακόμη και όταν εισέρχεται σε έδαφος Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διέπεται από ρωσικό δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, με στήριξη της νομικής της υπηρεσίας ισχυρίζεται ότι δεν θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Λέει όχι. Ακόμη και αν δεν εφαρμόσουμε την, την οδηγία για το φυσικό αέριο, υπάρχουν άγραφοι, ε, θυμοτυπικοί κανόνες δικαίου για την ενέργεια που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν μιλούμε, όταν μιλούμε για μια λειτουργία εξωχώρια ε, αγωγού όπως είναι ο θαλάσσιος Nord Stream 2. Θα πρέπει να υπάρχει αποσύνδεση από τον πάροχο, πρόσβαση των τρίτων μερών, μη διακριτικός προσδιορισμός των τιμών και διαφάνεια. Θα πρέπει αυτές οι, αυτοί οι άγραφοι κανόνες να ισχύουν και εδώ. Επιπλέον, ε, υπάρχει ανάγκη σύστασης ειδικού κανονιστικού καθεστώτος για τη λειτουργία του Nord Stream 2 που θα λαμβάνει υπόψη όλες αυτές τις προαναφερθήσεις αρχές και μάλιστα κάτι τέτοιο να γίνει μετά από διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, ζήτησε από το Συμβούλιο ή σύστησε στο Συμβούλιο, για να είμαστε πιο ακριβείς, σύστησε στο Συμβούλιο να αναθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κατάλληλη εντολή για τις σχετικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Στην ομάδα εργασίας για την ενέργεια της 28 Σεπτεμβρίου, η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου υπέβαλε την νομική γνωμάτευσή της, στην οποία δηλώνει ότι δεν είναι άμεσα εφαρμοστέα η οδηγία για το φυσικό αέριο, όπως σας είπα. Αυτό συμπίπτει και με τη, νομική, τη δική μας νομική υπηρεσία, τη γνωμοδότηση της δική μας νομικής υπηρεσίας, αλλά η γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου πάει πιο μακριά, γιατί ε, αρνείται την εφαρμογή των τεσσάρων αρχών που σας προανέφερα. Η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου θεωρεί ότι ε, αναπόκειται στην αμυγή πολιτική ε, ευχέρεια του Συμβουλίου αν κρίνει σκόπιμη μια τέτοια συμφωνία με τη Ρωσία για να εξασφαλίσει την ασφάλεια του ανεφοδιασμού και τη λειτουργία της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς. Αυτά τα δύο στοιχεία ε, περιχαρακώνονται στο άρθρο 194 της συνθήκης. Και εδώ ερχόμαστε στην πολιτική αξιολόγηση των κρατών μελών, στην πολιτική εκτίμηση. Πιστεύουν τα κράτη-μέλη ότι με την κατασκευή και τη λειτουργία αυτού του ε, αγωγού φυσικού αερίου ε, διακυβεύονται οι προαναφερθήσεις αρχές. Και αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να δοθεί σχετική εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για μας είναι λίγο φαϊνότερο βέβαια ότι υπάρχει ανάγκη θέσπισης ειδικού ρυθμιστικού πλαισίου στην περίπτωση αυτή για τους λόγους που σας εξήγησα. Τώρα, ο πρόεδρος ρώτησε πώς έχει η κατάσταση στο Συμβούλιο. Μέχρι στιγμής ε, δεν υπάρχει σαφής θέση υπό το φως και της νομικής γνωμάτευσης ε, της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου, γιατί αυτή η γνωμάτευση θα συζητηθεί μόλις μόνο αύριο, όπως είπε ο Πρόεδρος, στη νέα συνεδρία της Ομάδας Εργασίας για την Ενέργεια στο Συμβούλιο. Προς το παρόν πάντως, ε, διαπιστώσαμε ότι κάποια κρατημέλη είναι υπέρ της ανάθεσης εντολής. Για παράδειγμα, 7-8 χώρες μέλη είναι υπέρ της εντολής. Βέβαια, Κάποιες χώρες δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί, παραμένουν ουδέτερες. Καμιά δωδεκαριά. Και έχουμε και άλλες χώρες που προς το παρόν είναι πιο επικριτικές ως προς την ανάθεση εντολής και φαντάζεστε ποιες είναι αυτές οι χώρες. Τώρα, επανέρχομαι στο θέμα της εντολής. Μετά από ανάλυση της γνωμάτευσης της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι άσχετα με το αν θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εντολή, θα πρέπει παρόλα αυτά κάτι να γίνει, κάτι να κάνουμε. Γιατί είναι απαράδεκτο, απαράδεκτο να μην έχουμε μία ε, σαφή, αποκρισταλωμένη και κοινή άποψη για το ρυθμιστικό, κανονιστικό πλαίσιο των εξωχώριων αγωγών όταν φτάνουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε και προτίθεται να θέσει ένα τέρμα στην ε, έλλειψη ασφάλειας δικαίου που υπάρχει για το θέμα αυτό και όσο νουπο, κατά πάσα πιθανότητα τον επόμενο μήνα, θα καταθέσει νομοθετική πρόταση με κοινού κανόνες για τους αγωγούς φυσικού αερίου που θα εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά. Θα τεθεί έτσι ένα τέρμα στη νομική αβεβαιότητα. Και όπως είπε ο Ζαν Κλωδιούκερ παραπέμπτοντας αυτή τη νομοθετική πρόταση, υπογράμμισε την προσδοκία του η σχετική νομοθετική πρόταση να εγκριθεί και να τεθεί σε εφαρμογή μέχρι τα τέλη του 2018 το αργότερο του τεστίν, Αυτό το αδιαφιλονίκητο πλέον πλαίσιο που θα υπάρχει από τη στιγμή που εγκριθεί η σχετική νομοθετική πρόταση θα είναι πια ένα αδιαφυσβήτητο νομοθετικό πλαίσιο κανονιστικό που θα ισχύει και για τον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2. Αυτά και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε απορίες σας. Κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστούμε πολύ. Η συζήτηση είναι πολύ σημαντική. Δεν είναι πρώτη φορά βέβαια που γίνεται τέτοια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι ε, πρέπει εδώ πέρα να θυμόμαστε αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι ότι εμείς κάναμε τρεις συζητήσεις στην Ολομέλεια για το ζήτημα αυτό και μία κρόαση μάλιστα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. αποκινούμε το κονσόρσιουμ για τον ε, αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2. Όλα τα συμπεράσματα στα οποία αναφέρθηκε τώρα ο Διευθυντής Μπόρχαρτ ε, είναι αυτά στα οποία καταλήξαμε και εμείς κατά τη διάρκεια των δικών μας συζητήσεων και υπήρχε μια σαφής πλειοψηφία των συναδέλφων οι οποίοι είχαν ε, ουσιαστικά τις ίδιες απόψεις με τον Διευθυντή και μάλιστα στην τελευταία συζήτηση που έγινε πριν από ένα μήνα το διαπιστώσαμε και αυτό εκ νέου. Στα μέσα Σεπτεμβρίου δηλαδή. Συζητήσαμε τότε το ίδιο ζήτημα και καταλήξαμε στα ίδια συμπεράσματα. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν συζητάμε μία εντολή να είναι ενημερωμένε όλε οι επιτροπέ του Κοινοβουλίου ότι υπήρχε ήδη μία ομοφωνία, μία σύγκληση απόψεων, ήδη από τι συζητήσει που γίνανε κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας. Ο κύριο Σοντάλγας πρώτο, εκπρόσωπος πολιτικής ομάδας. Thank ε. Σας ευχαριστώ πολύ παρουσίαση ήταν απόλυτα σαφή. Βλέπουμε πώς κινούνται τα πράγματα. Το ερώτημά μου είναι πολύ σύντομο θα έλεγα και γενικής φύσης. Θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε με περισσότερες λεπτομέρειες ποιε είναι οι διαφορές ανάμεσα στο Nord Stream 1 που ήδη και το φυσικό αγωγό Nord Stream 2. Ποια είναι ακριβώς η διαφορά, ποια διαφορετικά χαρακτηριστικά έχουν, ποιες είναι οι βασικές ε, διαφορές τους και πως έρχεται ο δεύτερος αγώνας να συμπληρώσει τον πρώτο. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Βέρνερ τώρα έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ, σα ευχαριστώ και για την αλλαγή απόψεων την οποία κάνουμε σήμερα, γιατί δεν πιστεύω ότι το Nord Stream 2 δεν αποτελεί πολιτικό έργο. Η πολιτική πάντα υπησέρχεται σε τέτοιου ε, τομεί. Δεν είναι μόνο ποτέ αμυγό ε, οικονομικά τα ζητήματα αυτά. Είναι ασφαλώ πάντα και πολιτικά. Έχω κάποιε ερωτήσει να κάνω. Καταρχά, ό,τι αφορά τη διαφοροποίηση. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα αποτελέσει σημαντικό ε, θέμα. Οι κατοχώρε σε σημαντικό εμπορικό εταίρο θα βγει εκτό. Αυτό θα είναι σημαντικό από γεωλογική άποψη και πώ θα προσαρμοστεί η κατάσταση σε ό,τι αφορά το Nord Stream 2. Δεύτερη ερώτηση. Το ρυθμιστικό πλαίσιο. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλή ιδέα. Και η διαπραγματευτική εντολή. Αν ε, περάσει, που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα γίνει, αλλά αυτό είναι καλό. Ερωτώ, όμως, πώς μπορούμε να δώσουμε κίνητρο σε τρίτες χώρες να προβούν σε συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί στην τελική ανάλυση δεν γνωρίζουν τι γίνεται και δεν, μάλλον δεν υποχρεούνται να το κάνουν, δεν υπόκεινται σε κοινωτικό δίκαιο και αυτό δεν ισχύει μόνο για την Gazprom αλλά και για άλλους φορείς και παράγοντες. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα άλλαγε η τοποθέτησή σα εναντί του Nord Stream 2. Προθυμιστικό πλαίσιο θεωρώ ότι θα ήταν καλό να υπάρξει, γιατί ουσιαστικά δεν θα ίσχυε μόνο με το Nord Stream 2, αλλά για όλους τους αγωγούς αερίου που θα καταλήγουν στην Ευρώπη και που προγραμματίζονται για το μέλλον. Άρα θεωρώ ότι θα ήταν θετικό να υπάρξει μια δικτύωση, ένα συνδυασμό όλων αυτών για να ιδωθούν όλα αυτά στο πλαίσιο της συνολική διαφοροποίησης. Αυτά. Λοιπόν, και μια ερώτηση έχω για την Ουκρανία. Υπάρχει κάποιος επένδυτης που θα ε, επέκτηνε αυτόν τον αγωγό προκειμένου να συνεχίσει η ροή αερίου και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Okay. Ο κύριος Κρασνοντέμσκι, επόμενος ομιλητής. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που τόσο δραστήρια ασχολείται με το θέμα αυτό και με τέτοια ενέργεια γιατί η οδηγία για το φυσικό αέριο θα ήταν η, σωστή απάντηση, αλλά επισημάνεται κάποια νομικά κενά. Βέβαια και εμείς συμφωνούμε ότι θα πρέπει να ισχύουν κάποιες αρχές και στην περίπτωση αυτή. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, πολλοί ευρωβουλευτές, ώστε το ζήτημα αυτό να διευθετηθεί το συντομότερο δυνατόν. Θα ήθελα να πω ένα μόνο πράγμα. Ε, η συνάδελφος είπε ότι έχει και πολιτική σημασία αυτό το θέμα. Ε, το Nord Stream 2 δεν αφορά μόνο την ε, ενεργειακή μας ασφάλεια ή γενικώ το θέμα της ενέργειας ή γενικώ την οικονομία. Κατά κάποιο τρόπο το Nord Stream 2 είναι ένα σύμβολο. Σύμβολο των διπλών μέτρων και σταθμών. Γιατί σε μερικές χώρες ένας από τους λόγους της ανόδου του ευρωσκεπτικισμού είναι πρωτοβουλία σαν το Nord Stream 2, που δεν είναι πρωτοβουλία μόνο της Gazprom, γιατί η Gazprom έχει Ευρωπαίους εταίρους. Γιατί χωρίς Ευρωπαίους εταίρους δεν θα ήταν δυνατή τέτοια επένδυση από τη Ρωσία. Και γνωρίζουμε σε ποια χώρα θα καταλήξει αυτός ο φυσικός αγωγός και τι τεράστιο ρόλο παίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η κοινή γνώμη είναι πεισμένη ότι ε, ναι μεν αυτή η χώρα είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης αλλά ε, ενώ τη Γερμανία φυσικά δεν γνωρίζουν όλοι και το διαπιστώνω αυτό σε συζητήσει με τους φοιτητέ μου η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη δεν είναι ενημερωμένη για αυτό το θέμα. Ακόμη και οι φοιτητέ μου μερικές φορές το αγνοούν. Και εδώ δεν πλήττεται μόνο η Ουκρανία, αλλά και πολλέ χώρε τη Ανατολική Ευρώπη. Το σχέδιο αυτό έχει τεράστια σημασία και για την Ουκρανία και για πολλέ χώρε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Τεράστια σημασία και για την ίδια την ευρωπαϊκή ιδέα. Μπορεί να φαίνεται κάπω πομπόδε αυτό που λέω, αλλά πραγματικά το πιστεύω και καλό θα ήταν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο που από κάθε άποψη αντιβαίνει σε αρχέ Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ η Ρεμπέκα äh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξή. Η επιχειρηματολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Αλλά για μένα και για την ομάδα μου το όλο θέμα αυτό των μοναδικών επενδύσεων στον τομέα της ε, ενέργειας θέτει και το άλλο θέμα πέρα από την διαφοροποίηση των εισαγωγών αλλά και το ζήτημα της απαλλαγής από τον ανθράκα σε ό,τι αφορά τα μεγάλα λοιπόν αυτά έργα για εισαγωγές από μονάδες που χρησιμοποιούν ορεικτά καύσιμα, θα πρέπει να δούμε πώς θα τηρήσουμε και τις υποσχέσεις ε, του Παρισιού για να απαλλάξουμε από τον ανθράκα την οικονομία μας. Και εδώ λοιπόν υπάρχει μια ενδογενής αντίφαση, το τονίζω. Κατά τα άλλα πιστεύω ότι η Γερμανία έχει τη φιλοδοξία να υπάρξει συνεργασία με τη Ρωσία για το project αυτό, αλλά αυτό προκάλεσε μεγάλη ζημιά, γιατί με τον τρόπο αυτό οι υπόλοιπε ιδέε για την διαφοροποίηση και για καταπολέμηση των μονοπωλίων προκάλεσαν προβληματική κατάσταση σήμερα. Υπάρχει λοιπόν δεσπιστία στα ευρωπαϊκά κράτη σήμερα, η οποία σε αυτό ακριβώς οφείλεται ότι βρέθηκαν πρώτα τελεσμένου νου. Γερμανία και Ρωσία, παρά το γεγονό ότι διευκρινίζεται ότι πρόκειται για οικονομικό και όχι πολιτικό έργο, αλλά η Ρωσία παρ' όλα αυτά και η Γερμανία εδώ και πολλά χρόνια επιδιώκουν να βρουν συμφωνία. Ενώ οι υπόλοιποι είναι απλοί παρατηρητέ ουσιαστικά. Είναι λοιπόν σημαντικό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραμείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άκαμπτη έναντι του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Γιατί υπάρχουν πολλά συμφέροντα που διακυβεύονται, αναφέρθηκε η Ουκρανία. Δεν είναι μόνο όμως θέμα της Ουκρανίας, υπάρχει και ευρωπαϊκό συμφέρον. Υπάρχει λοιπόν η ευρωπαϊκή προοπτική της ε, Ουκρανίας και το έργο αυτό το οποίο αναπτύσσεται ουσιαστικά τάσεται κατά των οικονομικών συμφέροντων και των ε, πολιτικών προοπτικών της Ουκρανίας και έτσι θα πρέπει να είναι και προς το δικό μας συμφέρον να προωθήσουμε την Ουκρανία οικονομικά. Να μην το ξεχάσουμε λοιπόν αυτό ως παράγοντα. Κάτι άλλο το οποίο εντελώς ακατανόητο το βρίσκω, γιατί στη χώρα μου, στη Γερμανία, υπάρχουν τόσο πολλοί πολιτικοί που δεν έχουν ούτε καν αμφιβολία σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της ε, Υπήρου. Και δεν μιλώ μόνο για την ε, ασφάλεια παροχής ε, ενέργειας, αλλά για την πραγματική ασφάλεια, όταν 80% δεσμευόμαστε σε ό,τι αφορά τις αγωγές αερίου με, μία, με έναν αγωγό. Και μόνο. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάρμψα, ε, Μόλι το ανέφερε. Γιατί εισάγουμε άνθρακα από τη ΣΥΠΑ, αν θέλουμε να αυξήσουμε την ενεργειακή ασφάλεια. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Nord Stream, της νορβηγικού αγωγού και το αγωγού μεταξύ Λιβύης και Ιταλίας. Πώς είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σημείο αυτό να επιλέγει μόνο μία οικονομική συμφωνία και να μην ενδιαφέρεται καθόλου για άλλες. Πρόκειται για μία ξεκάθαρα πολύ επιλεκτική προσέγγιση. Δεύτερη ερώτηση, Πρόεδρε. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάγκασε τη Βουλγαρία και τα κράτη της των Βαλκανίων να εγκαταλείψουν το σχέδιο του South Stream. Αν δεν δώσετε, αν δεν είναι κάποιο σωτική απάντηση, προφανώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα, υπάρχει κάτι που πάει στραβά, κάτι άλλο. Η Νότιος Ευρώπη θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες αυτές, αλλά μάλλον θα το φροντίσει αυτό τώρα πλέον ο τοπικός αγώνα. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Κάρινς παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σας ζητώ συγγνώμη, δεν μπόρεσα να ακούσω την αρχή της παρέμβασης του Διευθυντή. Καθυστέρησα λίγο να φτάσουμε, ενημέρωσα λίγο για τα όσα είπαν. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση όσον αφορά το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με το φυσικό αυτό αγωγό του Nord Stream 2 και σε σχέση με τα όσα είπε η Ρεμπέκα Harms. Ξέρετε ότι έχουμε τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ξεκάθαρη αυτή η στόχη. Μείωση της χρήσης του άνθρακα, απαλλαγή από τον άνθρακα, αύξηση του ταγωνισμού, ε, μείωση της εξάρτησης από μία μονοχώρα και το καθεξής. Και σίγουρα ο Nord Stream αντιβαίνει στο πνεύμα όλων αυτών των στόχων που εμείς προωθούμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και που προωθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Δεν τίθεται λοιπόν κανένα ερώτημα όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική για τον τομέα της ενέργειας. Σίγουρα ο αγωγός αυτός αντιτίθεται στους βασικούς αυτούς στόχους. Βλέπουμε όμως ότι σε διεθνή ύδατα κατασκευάζεται περισσότερο ο αγωγός αυτός, οπομένως τίθεται και ένα ζήτημα δικαιοδοσία Ευρωπαϊκή ή μη. Όταν ο, αυτός ο αγωγό φυσικού αερίου βγει από τα νερά και τελικά φτάσει στην ευρωπαϊκή επικράτεια και σε ευρωπαϊκό Έδαφο, τότε πώ και κατά ποιο τρόπο αρχίζει να ισχύει η κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά τον ανταγωνισμό, όσον αφορά την ενέργεια και το καθεξή. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το ακόλουθο. Εσεί, ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εργαστείτε στα πλαίσια του ενωσιακού δικαίου, δικαίου που εγκρίνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο. Ξέρετε ότι η νομοθεσία πάντα μπορεί να βελτιώνεται. Και έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή λείπει κάτι από την νομοθεσία μας. Κάτι που θα την έκανε λίγο πιο δικτική, αν θέλετε, λίγο πιο δυναμική γιατί όταν εγκρίναμε όλε αυτέ τι σχετικέ νομοθεσίε στι οποίε αναφέρθηκα, νομίζω ότι δεν είχαμε καθόλου λάβει υπόψη μα τέτοιε περιπτώσει αυτή που συζητάμε σήμερα. Εσεί έχετε πραγματικά εντοπίσει τι αλλαγέ θα μπορούσαν να γίνουν στη δική μα νομοθεσία. Θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να προοδεύσουμε περισσότερο με κάποια στοιχεία τη κοινωτική μα νομοθεσία. Και αν τελικά εγκριθούν τέτοιε βελτιώσει από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό επιτρέπει σε εσά, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να έχετε τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να αναλάβετε δράσει. Ε, και να το πω και λίγο πιο ομά, να στραφείτε κατά του αγωγού αυτού που στρέφεται κατά τη Ενεργειακή Ένωση Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποιο άλλο που θέλει να πάρει το λόγο. Να πω κι εγώ κάτι με τη σειρά μου και προς ενημέρωση κάτι που θα είναι πολύ σημαντικό για τη συζήτησή μας. Την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τους συντονιστές, ορισμένοι είναι ήδη παρόντες στην αίθουσα, καθώς επίσης και τον υποφαινόμενο, ότι η αναθεώρηση της οδηγίας που έχει να κάνει με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και πιο συγκεκριμένα οι διασυνδετές και οι διασυνδέσεις, τα μέσα διασύνδεσης με τρίτες χώρες είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τουλάχιστον προβλέπονται από τους 8-6 διασυνδετές τους οποίους επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελε να προχωρήσει με τη μέθοδο fast track όσο το δηλαδή πιο γρήγορα. Και το ζήτημα αυτό θα συστηθεί εκ νέου σήμερα στις 5 το απόγευμα. Σε 45 λεπτά δηλαδή. Το ερώτημά μου είναι το ακόλουθο προς τον Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πότε θα έχουμε εμεί την πρόταση αυτή επιτάπητος επισήμως εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί βλέπετε ότι είμαστε σχεδόν έτοιμοι από τη δική μας την πλευρά. Μα έτοιμη είναι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ δύσκολο για μένα τώρα επί του παρόντος να σας δώσω μια συγκεκριμένη ημερομηνία, πάντως προβλέπετε η δημοσιοποίηση της πρότασης αυτής, πάντως την περιμένουμε για το πρώτο ήμιση του Νοεμβρίου, αυτό μπορώ να σας πω. Αν μου το επιτρέπετε τώρα θα ήθελα να απαντήσω σε ερωτήσεις που έθεσαν οι συνάδελφοι. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες. Κύριε Σάλαγκα, πολύ έύστοχε ερωτήσεις σας. Ποια διαφορά μεταξύ Nord Stream 1 και Nord Stream 2 και για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλάβαμε δράση νωρίτερα για το Nord Stream 1. Θα πρέπει να κάνω μια ιστορική αναδρομή εδώ πέρα. Ο Nord Stream 1 ήταν ένα εγχείρημα το οποίο καλωσόρισε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για την εποχή εκείνη θεωρούσαμε ότι αποτελούσε ακρογωνία ολίθο προκειμένου να αυξήσουμε και να βελτιώσουμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Ωστόσο, το ζήτημα του νομικού πλαισίου είχε τεθεί και τότε σε σχέση με τον Nord Stream 1. Η βασική όμως ιδέα τότε ήταν ότι τουλάχιστον την εποχή εκείνη, τουλάχιστον εκείνη την περίοδο, η Ρωσική Ομοσπονδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κατέλεγαν σε ένα γενικό πλαίσιο υποδομών στα πλαίσια του οποίου θα είχαμε θέσει όλες τις βασικές αρχές που θα έπρεπε να τηρηθούν σε σχέση με όλους τους αγωγούς συμπεριλαμβανομένου του Nord Stream 1. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο Μάλλον δεν, δεν συνειδητοποίησα ποτέ για ποιο λόγο δεν έγινε αυτό το πράγμα. Αυτή η συμφωνία πλαίσιο για τις υποδομές ουδέποτε τελικά συνήφθη την ε, Ρωσία και όταν άρχισα να ασχολούμαι με τον ενεργειακό τομέα και με όλες αυτές τις ρωσικές υποθέσεις είχαμε αναφέρει πολύ συχνά την προτινόμενη αυτή συμφωνία αλλά δεν υπήρξε τελικά καμία εξέλιξη και ξέρετε μετά με την προσάρτηση της Κρυμαίας η όλη αυτή η πρωτοβουλία κατέρευσε. Πάντως προβλεπόταν η τέτοια συμφωνία στον αφορά τις υποδομές και προφανώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να έχει κινήσει τη διαδικασία επί παραβάση αλλά εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο θεωρούσαμε ότι η υποδομή αυτή θα μπορούσε να λειτουργήσει και θετικά και γι' αυτό το λόγο τελικά καταλήξαμε στην, κατάληξη, στην κατάσταση που έχουμε τώρα, αντιμετωπίζοντας εντελώς διαφορετικά το Nord Stream 2. Να απαντήσω τώρα στη μητρική μου γλώσσα, στην κυρία Βέρνερ και στην κυρία Χάρμς. Θα μιλήσω λοιπόν τη μητρική μου γλώσσα, τα γερμανικά, αν δεν τα έχω ξεχάσει ακόμα. Κυρία Βέρνερ, η Διαφοροποίηση ναι και η Ολλανδική παραγωγή στο Groningen υπαναχωρεί, ε, πάει πίσω. Και με την υποχώρηση της παραγωγής στη Βόρεια Θάλασσα θα δούμε και η παναχώρηση περίπου 35.000 ε, κυβικών μέτρων σε χώρο επίπεδο. Το Nord Stream 2, ρωτάτε, είναι καλό στοιχείο στο πλαίσιο αυτό. Καταρχά, θεωρούμε ότι ένα μεγάλο τμήμα ή τουλάχιστον ένα μεγαλύτερο τμήμα των ποσών αυτών, των όγκων αυτών, θα ε, αντισταθμιστεί με εισαγωγή υγροποιημένου αερίου. του σχετικού όρου του δημιουργούμε τώρα. Όπω ξέρετε έχουμε τα τέρμιναλ τα οποία δεν έχουν επαρκέ σε υγροποιημένο αέριο και θα πρέπει και αυτά να μπουν πιο ε, δυναμικά στον ανταγωνισμό. Και οι αναλύσεις λοιπόν της Διεθνούς ε, Οργάνωσης Ενέργειας θεωρούν ότι θα διπλαστεί μέχρι το 2020 η εισαγωγή υγροποιημένου αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα ένα κομμάτι της απώλειας θα αντισταθμιστεί με αυτό. Ένα άλλο τμήμα φυσικά θα καλυφθεί και από ρωσικό αέριο, αλλά όχι μόνο από ρωσικό αέριο. Για παράδειγμα, περιμένουμε και αύξηση των εισαγωγών αερίου από τον χώρο της Μεσογείου, όπου έχουμε νέα κοιτάσματα στο Ισραήλ, στην Αίγυπτο δεν τίθεται μόνο θέμα ρωσικού αερίου. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μόνο το ρωσικό αέριο θα μας βάλει από την δύσκολη θέση και θα αντισταθμίσει ε, την υπαναχώρηση της εγχώριας παραγωγής. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Θέτεται μια πολύ καλή ερώτηση. Τι γίνεται γιατί εμεί ε, μόνοι μα ε, δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Ακόμα και αν λάβουμε την διαπραγματευτική εντολή, χρειαζόμαστε και την έγκριση και τη άλλη πλευρά. Προφανώ. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο αντιπρόεδρο Εύκοβιτ ε, συναντήθηκε με τον κύριο Νόβακ, τον Ρώσο ομόλογο του, και επέθεσε το θέμα αυτό. Ο Υπουργό Νόβακ, λοιπόν, ήταν ενδιαφέρον. Δεν είπε μόνο ότι «Α, κοιτάξτε, για μας τι μας νοιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο, δεν μας καλύπτει», αλλά ε, έδειξε διαλλακτικά. Διαλλακτική στάση είπε ότι παρακολουθούμε προσεκτικά τι ε, συζητήσει για την εντολή και αναλόγω θα λάβουμε και δική μα απόφαση. Νομίζω ότι αυτή η ε, προσεκτική στάση έχει να κάνει με το γεγονό ότι οι Ρώσοι γνωρίζουν πού βρισκόμαστε. Δεν είναι. Δεν θέλουμε να καταστρέψουμε οποιαδήποτε διαδικασία, απλά θέλουμε μια νομική βεβαιότητα και για του επενδυτέ. Άρα θεωρώ ότι όλοι οι συμμετέχοντες παράγοντες έχουν συμφέρον να τηρούνται οι υφιστάμενες ρυθμίσεις. Ναι, ρυθμιστικό πλαίσιο για όλους, προφανώς, προφανώς. Ναι, δεν είναι λέξη Gazprom, δεν είναι μόνο για το Gazprom ή μόνο για το Nord Stream 2 αυτή η νομοθεσία, προφανώς, αλλά θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι κάθε αγωγός πρέπει να ελέγχεται υπό τους συγκεκριμένου ξεχωριστούς του όρους. Τελευταία ερώτηση. Ουκρανία. Και τι γίνεται με τους αγωγούς ε, στην ε, Ουκρανία, κατά πόσον υπάρχουν επενδυτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια ομάδα εργασία με διάφορους φορείς και διαχειριστές ε, δικτύων στην Ουκρανία. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν λάβαμε σχετικά αποτελέσματα και πορίσματα και έτσι έχουμε την εξή αποστολή με την ε, Ουκρανική κυβέρνηση να διαπραγματευτούμε για το πώ θα διαμορφωθεί το συνολικό πακέτο αποσύνδεση σε ό,τι αφορά του φορεί και του διαχειριστέ, του και του διαχειριστέ των δικτύων. Δεν μπορώ να αναφέρω ονόματα, αλλά έχουμε τέσσερι ε, ε, ευρωπαϊκέ επιχειρήσει που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον προκειμένου να αναλάβουν να λάβουν μέρα, μέρος στο δίκτυο διανομής. Αυτό λοιπόν αποτελεί ένα πολύ μεγάλο επιχείρημα σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους, σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη διαμετακόμιση μέσω Ουκρανίας, αν υπάρχει τέτοια διαχείριση από αυτές τις επιχειρήσεις. Κυρία Χάρμς τώρα, θέτεται ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο μελλοντικές επενδύσεις. Γιατί εξακολουθούμε να επενδύουμε σε υποδομέ αερίου. Και αυτό δεν αφορά μόνο το Nord Stream 2, αλλά όλε τι υπόλοιπε υποδομέ Έχετε πάρα πολύ δίκιο, ξέρετε, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να αλλάξει τον τρόπο σκέψης της σε ό,τι αφορά την κατασκευή οποιαδήποτε καινούργιου αγωγού θα πρέπει να κοιτάξουμε κατά πόσο δεν μπορεί να γίνει βελτιστοποίηση των ήδη φυστάμενων αγωγών και η ψηφιοποίηση, γιατί μόλι ακούσατε την Επίτροπο για την ψηφιοποίηση, θα μα δώσει ακριβώ την ευκαιρία αυτή να επιφέρουμε μια βελτιστοποίηση τέτοια σε ό,τι αφορά την απαλλαγή από τον άνθρακα τώρα. Αυτό προφανώς συνδέεται με τον Nord Stream 2. Πρέπει να κάνουμε τη συζήτηση αυτή, γιατί αν πιστεύουμε στην ε, ηλεκτρική ενέργεια για όλους τους τομείς, ότι υπάρχει μόνο ένας κόσμος, ο ηλεκτρικός κόσμος, ή πιστεύουμε ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα χρειαστούμε ένα διπλό, διτό σύστημα, όπου δεν μπορούμε να καταργήσουμε εντελώς το αέριο, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αποχωρεί αυτή η τεχνολογία, αλλά Πρέπει να σας διευκρινίσω ότι έχουμε ήδη ένα εκτενέστατο δίκτυο εκτενή υποδομή το γεγονός. Η ερώτηση λοιπόν του κατά πόσον θα πρέπει να προωθήσουμε το ανανεώσιμο αέριο είναι κάτι το πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό θα το εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο επισταμένος. Θα προσπαθήσουμε και εδώ Ενδεχομένω να κάνουμε μια πιο εντελεχή σχετική συζήτηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ουκρανία και είπατε ότι είναι οικονομικό παραγοντά, προφανώ. Προφανώ. και θα ισχύει αυτό και στο μέλλον. Και τώρα να μιλήσω πάλι αγγλικά. Και να απαντήσω στον κύριο Κρασνοντεύσκη, τον καθηγητή Κρασνοντεύσκη. Δεν ε, ήταν ε, σαφώς ερώτημα αυτό το οποίο θέσατε, αλλά καταλαβαίνω την παρατήρησή σας. Οι πληροφορίες που έχουμε για όλα αυτά τα projects υποδομών είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και όντως ε, πρέπει να σας πω ότι υπήρχε ένα θετικό αφήγημα, θέλετε, και γύρω από τον, φυσικό, από τον αγώνα αυτό φυσικού αερίου. Ότι οι δυτικέ αγορέ καταναλώνουν 80% και από οικονομική πλευρά θα μπορούσε να υποστηρίξει κανεί ότι να φτάσουν άμεσα να φτάσει άμεσα το φυσικό αέριο εκεί πέρα που πραγματικά καταναλώνεται δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να επικρίνουμε αλλά όπως υπόθηκε και από κάποιους συναδέλφους σας και το είπα και εγώ πριν από λίγο, σε σχέση με τους στόχους πολιτικής που έχουμε στα πλαίσια της Ένωσης Ενέργειας, σε σχέση με το πνεύμα που υπάρχει στην Ενεργειακή Ένωση, δεν μπορούμε ουσιαστικά εμεί να αποδεχθούμε τέτοια επιχειρήματα με τέτοια προσέγγιση. Κύριε Κόχλιτσεκ τώρα. Είπατε ότι πολλές φορές είναι επιλεκτική η προσέγγισή μας. Δεν μπορώ να συμφωνήσω όμως μαζί σας. Δεν είναι επιλεκτική η προσέγγισή μας. Αναφερθήκατε εσείς στους αγωγούς της Νορβηγίας, του νορβικό αγωγό, νορβηγικό αγωγό. Μα αυτός καλύπτεται από διακυβερνητικές συμφωνίες οι οποίες συνήφθησαν μεταξύ της Γερμανίας και της Νορβηγίας. Εμείς αυτό το οποίο ζητάμε εδώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η διακυβερνητική αυτή συμφωνία να μπορούσε να ισχύει και προκειμένου. Αρχικά είχαμε πει στη Γερμανία κάντε το ίδιο πράγμα με το Nord Stream 2 και η γερμανική κυβέρνηση μα είπε α, όχι, όχι, εμεί δεν θέλουμε να πραγματευτούμε για αυτόν τον αγωγό. Επομένως το μπαλάκι επέστρεψε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρετε ότι ε, μπορεί διαπραγμάτευση να γίνει από κράτος μέλος προς τρίτη χώρα ή να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν αντιλαμβάνει η Γερμανία την ευθύνη αυτή, άρα πρέπει να το κάνουμε εμείς. Δεν είναι επιλεκτική προσέγγισή μας. Αλλά και οι αγωγοί αυτοί που έρχονται από την Αλγερία. Μα και σε αυτούς έχουμε συμφωνίες με τρίτες χώρες. Επομένως δεν παραβλέπουμε. Ξέρετε ότι η μόνη εξαίρεση είναι ο Nord Stream 1, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα πλαίσια ενός νομικού κενού ακόμα και σήμερα. Έπειτα, όσον αφορά τον αγωγό South Stream, μας ρωτήσατε για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάγκασε την ε, Βουλγαρία να εγκαταλείψει αυτή την πρωτοβουλία. Εμείς δεν κάναμε τίποτα τέτοιο. Ο λόγος για τον οποίο δεν ευωδόθηκε τελικά το South Stream είναι επειδή λήφθηκε μια απόφαση από τη ρωσική πλευρά. Εμείς αυτό το οποίο κάναμε ήταν να εφαρμόσουμε τους κανόνες που έχουμε για τις κυβερνητικές προμήθειες. Γιατί το Δεκέμβριο στη Βουλγαρία, όταν έγινε ένας δημόσιο διαγωνισμό από τις 23 Δεκεμβρίου μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, δηλαδή μετά τα Ορθόδοξα Χριστούγεννα, μόνο οι ρωσικές εφημερίδες ήταν αυτές οι οποίες δημοσίευσαν την προκήρυξη του διαγωνισμού. Αυτό επέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπε ότι πρόκειται για μια διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού, δημόσιων προμηθειών, η οποία τελικά παραβιάζει τους κοινοτικούς κανόνες. Και είπαμε ότι η προσέγγιση αυτή, η τακτική αυτή είναι απαράδεκτη και εν συνεχεία η Gazprom είπε «Α, εγώ εγκαταλείπω τώρα το South Stream και δεν δίνω συνέχεια στην πρωτοβουλία αυτή». Δεν πήρε την απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σίγουρα είχαμε προβλήματα με τον South Stream, αληθεύει αυτό, αλλά βρισκόμασταν σε φάση συζητήσεων με τη ρωσική πλευρά προκειμένου να καταλήξουμε στην αριθμιστικό πλαίσιο. Σας το λέω αυτό γιατί συμμετείχα προσωπικά σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αλλά επαναλαμβάνω, σταμάτησαν από τη δική μας πλευρά οι διαπραγματεύσεις τη στιγμή που η Ρωσία προσάρτησε την Κρυμαία και τότε τελείωσαν τα πάντα. Δεν αληθεύει πάντως ότι εμείς ε, αναγκάσαμε την Βουλγαρία να εγκαταλείψει το σχέδιο αυτό για τον South Stream. Τέλος κύριε Κάρντς. Πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Αυτό το οποίο θέτουμε επιτάπητο τώρα ως μελλοντική νομοθετική πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι να έχουμε μια πλήρη εφαρμογή της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια. Αυτή είναι τώρα η πρόθεσή μας με τις ε, τροποποιήσεις ε, που προβλέπουμε στα πλαίσια της οδηγίας για το φυσικό αέριο. Αλλά το βασικό ερώτημα είναι αυτό το οποίο θέσετε εν συνεχεία. Αρκεί αυτό θα είναι από μόνο το αποτελεσματικό. Αυτό μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι η πιο αποτελεσματική ριζοσπαστική αν θέλετε εξέλιξη θα ήταν να έχουμε βέτο τελικά. Να γίνει ένας πρώτος έλεγχος και έπειτα να δούμε τελικά αν το σχέδιο αυτό ευθυγραμμίζεται με τις δικές μας τις διατάξεις και τις πρακτικές. Πρέπει να δούμε τη συνεχεία πώς θα τοποθετηθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Ξέρετε ότι σε περίπτωση βέτο θα είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να δικαιολογήσουμε τη στάση αυτή, τουλάχιστον στα διεθνή φόρα στα οποία συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή θα είναι η πραγματική πρόκληση, το να εφαρμόσουμε την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια είναι κάτι το οποίο τελικά θα μας βοηθήσει, θα μας διευκολύνει να καταφέρνουμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα όλους αυτούς τους αγωγούς φυσικών αερίων, γιατί θα έχουμε και καλύτερο ανταγωνισμό αλλά και υψηλότερο βαθμό διαφάνειας. Η τιμολόγηση επίσης ε, θα διαμορφωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα αρκεί όμως αυτό από μόνο του, αμφιβάλλω, γιατί φαντάζομαι ότι θα προκύπτουν και νέοι αγωγοί όπως ο Nord Stream 2 για παράδειγμα που μπορεί μεν να συνάδει με τις αρχές αυτές που θέτει δηλαδή η ευρωπαϊκή πλευρά αλλά τα βασικά προβλήματα που έχουμε σε σχέση με τους στόχους πολιτικής θα εξακολουθούν να υφίστανται ακόμα και αν καταφέρουμε τελικά να κάνουμε τον αγωγό αυτό να συμμορφώνεται με την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια, πάλι θα υπάρχουν βασικές θεμελιώδεις διαφορές όσον αφορά τους βασικούς στόχους πολιτικής που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να διασκεδάσουμε τα προβλήματα αυτά εφαρμόζοντας απλώς και μόνο την τρίτη δέσμη μέτρων. Δεν λέω ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε τη διαδικασία fast track. Για το 2020 έχουμε θέσει ως στόχο να έχουμε μία πλήρη πρόταση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το φυσικό αέριο που θα περιλαμβάνει πολλά από τα πράγματα που σας παρουσίασα σήμερα. Και ενδεχομένω να πρέπει να, να εξετάσουμε εκ νέου την πρόταση αυτή και να δούμε εν συνεχεία αν ε, ένα ενδεχόμενο βέτο έπειτα μπορεί να υποστηριχθεί από μας στα πλαίσια της ε, των διεθνών οργανισμών στους οποίους συμμετέχουμε, γιατί θεωρώ ότι μόνο τελικά με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε τα προβλήματα τα οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή με τον Nord Stream 2 και με αντίστοιχους αγωγούς. Σας ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά για τις απαντήσεις σας και τις παρατηρήσεις σας. Μας έχει απομείνει λίγη ώρα. Οπότε να θέσω και άλλες ερωτήσεις, άμα επιτρέπετε. Ή μάλλον να δώσω το λόγο στον κύριο Λάγκεν. Ναι, δυστυχώς καθυστέρησα γιατί ε, στο πρόγραμμα έλεγε μέχρι 4 η ώρα η επιτροπη σε πάση περιπτώσει. Σας ζητώ συγγνώμη αν θα θέσω ερωτήματα τα οποία ήδη έχετε ακούσει. Καταρχάς για την νομική βάση για το άρθρο 94, δεν θα υπάρξει σχετική γνωμοδότηση και πώς μπορούμε να καταφέρουμε το Συμβούλιο να λάβει αποτελεσματικά αποφάσεις. Μία ερώτηση επίσης, πέρα από το δικαίωμα βέτου το οποίο αναφέρεται, πώς θα διαμορφωθεί τα πράγματα. Και μία ερώτηση ακόμα, ίσως το έχετε αναφέρει, δεύτερη λοιπόν ερώτηση, αν σωστά κατάλαβα. Η νομική βάση ήταν σαφή για τον Nord 1 και δύο Είπατε ότι είναι η επιθυμητή υποδομή συμμετέχουν τα κράτη-μέλη στα πλαίσια της διαδικασία της περιβαλλοντικής και το καθεξής και είπατε μεταξύ Γερμανίας και Νορβηγίας υπήρξε διμερή συμφωνία. Αν λοιπόν η Γερμανία με τη Ρωσία συνεχί... λάμβει ε, και καταλήξει σε συμφωνία με τη Ρωσία η καγκελάριος είναι υπεύθυνη για αυτά. Αυτό επαρκεί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως νομική βάση. Στέκει αυτό. Και μπορείτε να μας πείτε γιατί η Γερμανία ως τώρα ήταν αντιστακτική και κατά πόσον είναι η συνδυσμένη διαδικασία που η Γερμανία ουσιαστικά παίρνει απόφαση μόλι την έχουν πάρει και οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση follow-up, επιτρέψτε με μία περώτηση. Άκουσα αυτά που είπατε και ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Αυτό που λέτε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούσε θα μπορούσε να προβάλλει βέτο, αλλά μπορεί να μην σταθεί αυτό στα πλαίσια του ΠΟΕ. Εγώ σκέφτομαι αυτή τη στιγμή ως ε, υπερασπιστής των, ε, των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Μπορούμε να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε και ενδεχομένω να αποφασίσουμε να μην προβάλλουμε βέτο εάν δεν γίνει σεβαστό. Αλλά στην περίπτωση αυτή μπορεί να παραβιαστούν αρκετά ζητήματα σε ό,τι αφορά τον upstream. Άλλο τρόπο θα ήταν να υποβληθεί το βέτο, να περάσει στο ΠΟΕ το θέμα αυτό και ενδεχομένω αυτό να έχει πιο πολλά αποτελέσματα. Γιατί στον ΠΟΕ να έχουμε οι πιθανότητε να νικήσουμε. Γιατί αν δεν έχουμε προσπαθήσει, πώ θα ξέρουμε αν θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε. Γιατί να μην ε, τροποποιήσουμε λοιπόν την νομοθεσία και λοιπόν, να μην υποβάλουμε βέτο. Τι έχουμε να χάσουμε, γιατί αν δεν πάμε καν στον ΠΟΕ, θα έχουμε ήδη χάσει, θα είμαστε ήδη χαμένοι σύμφωνα με αυτό που μας είπατε. Κύριε Μπορχαρτ, άλλες δύο ερωτήσεις επιτρέπεστε μου, κύριε Σκόχκλητσέκ. Όταν ήταν εδώ η Ουκρανική Αντιπροσωπεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας ε, ανέφεραν ότι ο αγωγός αυτός, όπως είπατε, είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Φανταστική, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει τεχνικός πώς. Δεύτερη ερώτηση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φροντίζει τη δικτύωση των αγωγών αερίων μεταξύ ε, Νότου και Βορρά. Υπάρχουν σχετικές αποφάσεις και θα μπορούσε να έχει γίνει, να έχει ολοκληρωθεί αυτό. Ωστόσο δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί, γιατί δεν ε, εξασφαλίσατε την παροχή αερίου της στην, στην Νότια Ευρώπη από, άλλους, ε, από πηγές, από την Τουρκία, τον Αμπούκο ή με Ρώσους, Βούλγαρους στο South Stream. Και γιατί δεν ετέθησε καμία ερώτηση για το Ιράν. Το Ιράν έχει τεράστιες δυνατότητες εξαγωγής φυσικού αερίου. Τα τα ξέρετε όλα αυτά βέβαια. Uh, Σας ευχαριστώ. Άλλος κανείς παρακαλώ θέλει το λόγο για να υποβάλει ερωτήσεις, γιατί τρίτος γύρος δεν πρόκειται να γίνει. Όχι, ουδής άλλος, οπότε ο διευθυντής ο κύριος Μπόρχαρτ έχει το λόγο. Κύριε Λάγκε. Επιβεβαιώνω. Η νομική βάση θα είναι το άρθρο 194 της συνθήκης. Και με βάση αυτό το άρθρο θα προωθήσουμε την πρότασή μας. Ρωτήσατε γιατί η Γερμανία δεν ξεκίνησε διμερείς συζητήσεις με τη Ρωσία. Ειλικρινά δεν γνωρίζω, ομολογώ ότι δεν το ξέρω αυτό. Και ε, θέσαμε την ερώτηση σε όλα τα επίπεδα. Επιτροπής, Αντιπροέδρου, η μόνη απάντηση που λάβαμε είναι ότι δεν είναι απαραίτητο, δεν χρειάζεται διμερής επαφή. Οπότε, οχυρώθηκαν πήρα από τη, νομική υπηρεσία, τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας ότι δεν είναι εφαρμοστέο το ενεργειακό δίκαιο και άρα δεν χρειάζεται καμία διαπραγμάτευση. Αυτή είναι η μόνη εξήγηση που έλαβα. Βέβαια, η Γερμανία εξακολουθεί να επιμένει σε αυτή τη θέση στην ομάδα εργασία του Συμβουλίου. Οπότε στο μέτωπο αυτό έχουμε τις ε, συνέπειες. Κύριε Κάρης, καλή ιδέα σα Δίκιο έχετε ότι όποιος την ε, ε, διερεύνηση και αυτή της πιθανότητας με σοβαρό τρόπο, αλλά όχι εσπευσμένα ή βεβαιασμένα. Θα πρέπει πρώτα να εκπονήσουμε μελέτη αντικτύπου και αυτή η διαδικασία είναι πιο χρονοβόρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πιο fast track διαδικασία για να καταστήσει εφαρμοστέο το ε, τρίτο πακέτο, τρίτη δεσμή για την ενέργεια. Το θέμα είναι αρκεί αυτό ή θέλει, χρειάζονται και κάποιες επιπλέον ενέργειες. Κύριε Κόχλιτσεκ, όταν βλέπουμε τις άλλες, τους άλλους αγωγούς, τι να σου πω, ποια είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι αν πάρετε τον αγωγό δια, διαμετακόμισης, είναι 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια, αμερικανικά δολάρια, γιατί είναι δύο η αγωγή. Δεν είναι ότι έχει καταστραφεί, αλλά ο Γιούκα, η Γιούκα Τρασγκάς, αυτός ο όμιλος, δεν έκανε το καθήκον του και δεν επανεπένδυσε τα τέλη διαμετακόμισης στη συντήρηση, τον εξυγχρονισμό του συστήματος. Πρέπει να γίνουν κάποιες επενδύσεις, αλλά όχι τα 12 δισεκατομμύρια που ισχυρίζεται η Gazprom, τα 12 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια. Εμείς ε, έχουμε πληροφορίες για πολύ χαμηλότερο ποσό επενδύσεων που χρειάζεται. Τώρα για τον South ε, Stream ή τον Αμπούκο ή ε, άλλη αγωγή του νότιου διαδρόμου δεν αποκλείονται. Έχουμε ε, από το Connecting Europe Facility τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Αυστρία. Αυτό το διάδρομο σε μεγάλο βαθμό ακολουθεί την πορεία του Ναμπούκο η, η πρωτοβουλία αυτή. Και αναφερθήκατε και στο Turk Stream. περιμένουμε και το Turk Stream 1 και θα φέρει ε, ταχύτατα φυσικό αέριο από τη Ρωσία στην Τουρκία. Το θέμα είναι το Turk 2, αν θα εφαρμοστεί και τι θα γίνει με αυτό. Εδώ οι πληροφορίες μας από τη Ρωσία είναι ε, αντιφατικές. Λένε ότι έχουν πουλήσει αέριο από την Ελλάδα στην Ιταλία. Το ίδιο το αέριο το υποσχέθηκαν όμως και στην Βουλγαρία μέσω διαμετακόμισης. Και πραγματικά δεν ξέρει κανείς τα πραγματικά σχέδια της Gazprom. Γιατί πετάνε στο τραπέζι πολλές και διάφορες ιδέες, προσπαθώντας να διχάσουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, δίνοντας λίγα πλεονεκτήματα στον καθένα, προσπαθώντας να διαταράξουν την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα για τη Βουλγαρία και το South Stream. Όταν οι Ρώσοι κατήργησαν το South Stream, γιατί δεν φταίμε εμείς, οι Ρώσοι το ανέρεσαν, ο Πρωθυπουργός Μπόρισοφ της Βουλγαρίας παραπονέθηκε και είπε και τώρα τι να κάνω εγώ. Ε, οπότε αναπτύξαμε ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με τη βουλγαρική κυβέρνηση για το Balkan Gas Hub. Ε, είπαμε στη Βάρα να δημιουργήσουμε ένα κόμβο, μια πλατφόρμα ε, συναλλαγών για να εξασφαλίσουμε φυσικό αέριο σε όλη την περιοχή, όχι μόνο φυσικό αέριο από αγωγό, αλλά και από το τερματικό υγροποιημένο φυσικό αέριο της Ελλάδας, ώστε να έχουμε γραμμή διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, Βουλγαρίας και Σερβίας και ήδη έχουμε αναθέσει μια γραμμή διασύνδεσης μεταξύ Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Οπότε, στο μέτρο θα έχουμε πλέξει γκάς από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Και αυτό θέλουμε. Θέλουμε να δημιουργήσουμε οικονομική αξία στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Να μην αφήσουμε την νοτιοανατολική Ευρώπη ε, εξαρτημένη από τους δυτικούς κόμβους αερίου. Θέλουμε και στην νοτιοανατολική περιοχή να αναπτύξουμε κόμβους για διαφοροποίηση, γιατί μέχρι στιγμής ε, εξαρτώνται πλήρως από το ρωσικό φυσικό αέριο, κάτι που δεν είναι βιώσιμο. Γι' αυτό και θέλουμε να δημιουργήσουμε τέτοιες πλατφόρμες. Οπότε είμαστε πολύ πιο διορατικοί ε, και πολύ πιο προχωρημένοι και στη σκέψη μας ε, και στα έργα μας από ό,τι πιστεύετε κύριε Κόχλησεκ. Σας ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά για την παρουσία σας, για τις ε, διεξοδικές πληροφορίες που μας δώσατε, για τη σχολαστική απάντηση σε ερωτήσεις, την καρποφόρα συζήτηση και περιμένουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Πολύ σημαντική ενημέρωση πάντως. Ε, σας ευχαριστώ. Έχουμε συνεδρίσει των συντονιστών σε μισή ώρα, οπότε σας αποχαιρετώ. Περνάμε στο τελευταίο σημείο της ε, δημόσιας συνεδρίασής μας. Την ενημέρωση από την ε, αποστολή της Επιτροπής Ήτρες στην Πολωνία. Είχαμε μία ολιγομελή ομάδα. Μπόνι, Σπυράκη, Βιμπάτσκα, Κρασνοντέμσκι και ε, μεταξύ 22 και 23 Μαΐου 2017 μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ήτρε επισκέφθηκε την Πολωνία σε διαρευνητική αποστολή ως προς τις αρμοδιότητες της Ήτρε. Όπως σας είπα, τα μέλη της αντιπροσωπείας ήταν ε, αυτά που σας προανέφερα και τα κίνητα της αποστολής ήταν τρία. Καταρχήν, να ενημερωθούμε καλύτερα για το ενεργειακό μείγμα τη Πολωνίας και για τις καινοτομίες στον τομέα τη καθαρής ενέργειας. Συνάντηση με ιδρυτές και επιχειρηματίες συναφιών επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιληφθούμε από πρώτο χέρι την καινοτόμο του προσέγγιση και τι προκλήσει που αντιμετωπίζουν. Και τρίτο κίνητρο να διαμορφώσουμε καλύτερη ιδέα για τον αντίκτυπο που έχουν τα κοινοτικά κονδύλια σε αυτούς τους κλάδους και πώς η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί. Η αντιπροσωπεία μας επισκέφθηκε τη Βαρσοβία και Κρακοβία. Είχαμε ένα υπερπλήρες πρόγραμμα συναντήσεων με πολλούς ε, συμφεροντούχους, πολλούς και διάφορους. Την πρώτη μέρα στη Βαρσοβία συναντήσαμε πολλές καινοτόμες νεοφύης επιχειρήσεις ε, που ενεργοποιούνται σε, στην προσφορά ψηφιακών λύσεων για την ηλεκτρονική υγεία και κάποιες νεοφύης επιχειρήσεις από τον ψηφιακό κλάδο. Επίσης, επισκεφτήκαμε το Campus Warsaw, το τεχνολογικό κέντρο ICM και το κέντρο δημιουργικότητας Ταργόβα 56. Εκεί μας υποδέχθηκε ε, ο αντιδήμαρχος της Βαρσοβίας. Πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη, ε, γιατί το κέντρο ήταν κάτι παραπάνω από κέντρο δημιουργικότητας. Μας υποδέχτηκε ο αντιδήμαρχος της Βαρσοβίας, ο κύριος Ολσεύσκη. Και την τελευταία μέρα μεταβήκαμε, τη δεύτερη μέρα μεταβήκαμε στο Ζάμψε, σε ένα κέντρο καθαρής τεχνολογίας άνθρακα και κατόπιν πήγαμε στην Κρακοβία για μια ευρυθή επίσκεψη του τεχνολογικού πάρκου ε, της Κρακοβίας και του ε, Κέντρου Επιστημών της Ζωής της Κρακοβίας. Επίσης συγκεντρώσαμε πολύτερες πληροφορίες από πρώτο χέρι που θα μας ε, εμπλουτίσουν τις συζητήσεις και την εκπόνηση νομοθετικών εκθέσεων στο μέλλον και θα βελτιώσουμε και έτσι και το έργο της Επιτροπής μας. Και μια ενδιαφέρουσα, ένα μυστική φωτογραφία από, τις, από την επίσκεψή μας αυτή στην Πολωνία. Αν τη θέλετε, μπορούμε να σας τη στείλουμε αυτή τη φωτογραφία. Θέλει κάποιος από τα μέλη της αντιπροσωπείας να προσθέσει κάτι στην ενημέρωση που έκανα. Όχι. Άλλος κανείς. Όχι. Παρατηρήσει σχόλια. Τίποτα άλλο. Όχι. Οπότε ολοκληρώσαμε και την ε, απογευματινή μας συνεδρία σε τη δημόσια και στις 5 σε 19 δηλαδή λεπτά θα συνεδριάσουν ξανά και σε λίγο μάλλον οι συντονιστές. Η υπόλοιπη επιτροπή αύριο το πρωί στις 9 με ένα πλούσιο πρόγραμμα που θα διαρκέσει μέχρι τις 12.30 από ό,τι ξέρω. Αύριο θα ολοκληρώσουμε στις 12.30. Το αυριανό απόγευμα είναι ελεύθερο. Δεν έχουμε συνεδρίαση. Και ραντεβού με τους συντονιστές σε 18 λεπτά.